Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen, insbesondere diejenigen, die... Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας χαιρετήσω ιδιαίτερα εκείνους που δεν είδα σήμερα το πρωί. Συνεχίζουμε με πολύ πλήρη ημερησία διάταξη πάλι και θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω, να σας παρακαλέσω και όλους τους αδέλφους που ήρθαν τώρα να προσπαθήσουμε 20 λεπτά το πολύ να χρησιμοποιήσουμε για κάθε σημείο. Το πρώτο θέμα που έχουμε προς είναι το σημείο 11 της ημέρας της διάθεση, διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτώνων. Αρμόδιος τη χνομοδότηση είναι ο κ. Καρίν, που είναι παρόν. Και εξ αυτού θα ήθελα να δώσω και το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα που αναφέρατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος μεν, σαφής δε. Όπως λέω και στην γνωμοδότησή μου, προσπαθώ να τονίσω τα προβλήματα που θεωρώ ότι υπάρχουν στην τρέχουσα οδηγία. Είναι σημαντικό ο νέος κανονισμός που θα υπάρξει για τη διάθεση στην αγορά και χρήση των βιοκτώνων προϊόντων να βελτιώσει το σύστημα που ισχύει σήμερα. Στην απάντηση της, ε, της Επιτροπής ε, τονίστηκε ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια συγκεντρωτική ε, υπηρεσία επιπλέον από τις υπηρεσίες αδειοδότησης των κρατών μελών. Νομίζω ότι η αρχική πρόταση περιόριζε ιδιαίτερα την διαδικασία αυτή στην πολύ αυστηρή ταξινόμηση των χημικών ουσιών. Από την άλλη μεριά, δεν είναι νομίζω σωστό να διευρύνουμε ευρωπαϊκά μία ουσία που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι είναι καλά σε όλες τις χημικές ουσίες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε μία λειτουργούσα εναλλακτική, έχω προτείνει κάτι σχετικά με τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου, και επίσης η τελική οδηγία να μην υπάρχει από το 2023 αλλά από το 2016. Εάν αποδειχθεί καλή θα μπορεί να διευρυνθεί. Έχουμε όμως επίσης κατά ότι τα περισσότερο διοκτώνα προϊόντα θα εξακολουθούν να εγκρίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη και ότι η αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να βελτιωθεί γι' αυτό όπου είναι δυνατό. Ελπίζω ότι κάποια από τα μέτρα που προτείνω θα είναι σύμφωνα με το στόχο αυτό. Σε μία αγορά, κατά την οποία πολλοί συμμετέχοντες είναι ΜΜΕ, έχω προτείνει εθνικά γραφεία ενίσχυσης για να μπορέσουν να βοηθούν τις επιχειρήσεις αυτές πριν θέσουν το προϊόν τους στην αγορά. Προτείνω επίσης το τίσιο τέλος να μην εφαρμόζεται για τις ΜΜΕ που χρησιμοποιούν την ε, την κεντρική μάλλον διαδικασία ε, έγκρισης. Επίσης έχω προτείνει ομοιόμορφες προθεσμίες για να επιταχυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο μπορούν να δοθούν οι άδειες. Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, προτείνω ένα πιο απλούστερο σύστημα ε, για να μπορέσουν οι κεντρικές αρχές να εφαρμόζουν πιο αυστηρές, ε, αυστηρούς προϋποθέσεις, αν χρειάζεται. Όσον αφορά το πλαίσιο, θα ήθελα να προσπαθήσω να έχω πιο κεντρική, πιο γενική διατύπωση. Θα πρέπει δηλαδή να προτείνεται τα γενικά τεστ των ε, ενεργών ουσιών που αναφέρονται στο 5.1 γάμα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές με άλλη νομοθεσία. Είχαμε πολλές επαφές με λόμπι των ε, επιχειρήσεων και αναφέρεται ότι οι απαιτήσει για την αδειοδότηση να είναι μόνο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την ετικεθοσία. Θα υπάρχουν όμως οι σχετικές τροπολογίες 37 και 39 στην πρότασή μου για να παρουσιάσουμε τι θα γίνεται όταν υπάρχουν σε μία ένα κράτος μέλος περισσότερες στις μία επίσημες γλώσσες. Αυτά με δύο λόγια είναι τα κύρια σημεία που παρουσιάζω στην γνωμοδότησή μου. Καλό βέβαια τους συναδέλφους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Και όπου μπορώ θα προσπαθήσω να τις ενσωματώσω στην έκθεσή μου, εφόσον αυτό θα μας βοηθήσει να κινηθούμε προς μια θετική κατεύθυνση. Ο πρόσωπος της Κομισιόν είναι παρόν, είχε την καλοσύνη να μου συστηθεί και θα ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τις δικές του αντιδράσεις στα θέματα που παρουσίασα και βέβαια και στο γραπτό κείμενο που έχω υποβάλει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πατριτσέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Κάριμ για την εξαιρετική δουλειά του ε, και σε μεγάλο βαθμό συμπεριλαμβάνει και πολλές προτάσεις που είχα επιβάλει εγώ σε προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σήμερα η αγορά των βιοκτώνων φτάνει τα 890 εκατομμύρια αργό και το ένα μεγάλο μέρος της αγοράς αυτής ελέγχεται από τρεις μεγάλους ομίλους. Έτσι λοιπόν αυτός ο κανονισμός που θα τροποποιήσει την οδηγία του 98 θα πρέπει να εξισορροπήσει τα συμφέροντα μεταξύ των μεγάλων ομίλων και της εναρμόνισης με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γιατί η οδηγία γεννιόταν από βάση δύο στόχων προστασία της υγείας και προστασία του περιβάλλοντος και ε, εμφανίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια μία σειρά προβλημάτων και απαγορευτικό κόστος ε, προέκυψε. Έτσι λοιπόν υπήρξε μία σειρά προβλημάτων που σε κάποιο βαθμό η Κομισιόν προσπάθησε να ρυθμίσει με αυτόν τον κανονισμό που παρουσιάζεται σήμερα σε εμά. Έχουμε μια νέα εκδοχή λοιπόν της νομοθεσίας. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός ο κανονισμός αυτός ε, και παρουσιάζει μια σειρά προβλημάτων ε, σε εμά και πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εν γέννη. Το κείμενο της Κομισιόν είναι καλό θα ήθελα λοιπόν εγώ να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ε, στο κείμενο του εισηγητή ε, εγώ θα παρουσιάσω λοιπόν κάποιες τροπολογίες που ελπίζω ότι η Επιτροπή και οι συνάδελφοι ε, θα δεχτούν θετικά. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ορισμένες πτυχές του κανονισμού για τα βιοκτώνα που είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσες. Ε, από ό,τι κατάλαβα, ο εισηγητής ε, συμφωνεί με την αναγκαιότητα να υπάρχει κεντρική διαδικασία διοδότησης για τα βιοκτώνα με χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο όφελος, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και με τέτοιο βαθμό, έτσι μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Και επίσης συμφωνώ ε, απόλυτα με το ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο ε, για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αντιοδότηση. Επίσης, ε, όρος μειωμένο κόστος φαίνεται να είναι ειδικά, μάλλον να είναι αρκετά όριστος. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Έτσι λοιπόν θα προτείνω στην Επιτροπή κάποιες τροπολογίες για να καθοριστούν κριτήρια βάσει των οποίων θα έχουμε συγκεκριμένα ποσά που θα τίθενται ξεκάθαρα. Συμφωνώ με τον εισηγητή για την αναγκαιότητα να ε, μην καταβάλουν το ετήσιο τέλος η μία ε. Τώρα, σε ό,τι ε, αφορά τα εμπόδια και την αποφυγή τους, πιστεύω ότι να χρησιμοποιεί κανείς την επίσημη γλώσσα της χώρας του πρέπει να αρκεί για την αδειοδότηση να επενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν μεγαλύτερη αρρωγή στις επιχειρήσεις ε, προβλέποντας ε, βάσεις δεδομένων προκειμένου να μην δημιουργούνται επικαλύψεις ε, και να μην ζητούνται δύο φορές τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεπάζ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την ποιότητα της έκθεσής του και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που μου φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχήν, ε, ο ορισμός του μικρού κινδύνου. Τι εννοεί ο εισηγητής των διεύρυνση της κατηγορίας του μικρού κινδύνου, γιατί εγώ έχω πρόβλημα με τον ίδιο τον ορισμό και αν πρόκειται να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο θα ήθελα να ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. όσον αφορά την ε, εξάλληψη των επικινδύνων ουσιών. Εγώ συμφωνώ με ορισμένα κράτη-μέλη που λένε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οι, ουσίε οι ουσίες οι οποίες είναι ε, ιδιαίτερα δηλητηριώδεις και οι οποίες συγκεντρώνονται στον οργανισμό. Θα πρέπει να το ξάσουμε και αυτό. Τώρα, ετικέτες. Καταλαβαίνω ότι για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να είναι σωστά ενήμερος ο κατανοητής για το τι αγοράζει και δεν θα πρέπει να αποφύγουμε εκ μιας αρχής το θέμα της ετικετοθεσίας ή της σήμανσης. Κατόπιν, υπάρχει το θέμα της διεύλυσης της κοινωτικής διαδικασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Καταλαβαίνουμε βέβαια την ησυχία της βιομηχανίας για τη διαδικασία αυτή, η οποία είναι και δαπανήρη. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι έμεσες επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε σωστά το θέμα. Καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν το σύστημα γιατί υπάρχει κάποιο έσοδο από αυτό και με αυτό μπορεί να χρηματοδοθούν οι εθνικές έρευνες, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε κάποιο μέσο όρο. Ανησυχώ κάπως για το κείμενο που έχουμε μπροστά σχετικά με τις ΜΜΕ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο κείμενο που να καθιστά την πρόσβαση στην αγορά για τις ΜΜΕ αδύνατη. Ο εισηγητή ή ο προλαλή αναφέρθηκε στο ότι υπάρχουν τρει μεγάλε επιχειρήσει που καλύπτουν ε, το μεγαλύτερο ποσοστό του τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα οικονομικά στην αγορά και δεν θα πρέπει να αποτρέψουμε να παρεμποδίσουμε τις ΜΜΕ από την πρόσβαση του στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης το θέμα της πρόσβασης στα στοιχεία. Και αυτά που είπα για τις ΜΜΕ ήταν κάτι το οποίο οδηγήθηκα να αναφερθώ λόγω του γενικού θέματος. Αυτά με δύο λόγια κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας πω για το κείμενο που είναι ένα κείμενο που ίσως δεν κινητοποιεί πολλούς συναδέλφου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σπυρίλο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι τροπολογίε που προτείνονται από τον εισηγητή στην έκθεσή του μας βρίσκουν σύμφωνους ευρέως. Πολλές εξ αυτών ε, οδεύουν προς ε, την κατεύθυνση που επιθυμούσα και εγώ, δηλαδή να περιορίσουμε τις προθεσμίες για την απόκτηση της άδεια ε, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όμως, στο άρθρο 3 θα ήθελα να βάλουμε κάποιους ορισμούς όπως λόγω χάρη αυτής της δικηπητικής τροποποίησης ή τροποποίησης ε, μικρής οντότητας που προτείνονται στην πρόταση κανονισμού αλλά χωρίς να υπάρχει ένδειξη για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η ενσωμάτωση και πώς θα πρέπει να γίνει η ερμηνεία. Εδώ πρέπει να μην αφήσουμε δυνατότητα σε αποκλίνουσες ερμηνείες από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, του κανονισμού που πρέπει να διευκρινιστούν ή να εξηγήσουμε τι ακριβώς ε, λέμε όταν ε, λέμε συγκριτική αξιολόγηση των βιοκτώνων. Εκεί γίνεται αναφορά στο κείμενο της Επιτροπής, αλλά δεν αναφέρεται πώς πρέπει να γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρέμβουμε και εγώ σκέφτομαι να παρουσιάσω σχετικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση της αδειοδότησης, της άδειας, συμφωνα με το το άρθρο 24.1, η αίτηση πρέπει να γίνεται 18 μήνες πριν, 12 ε, μήνες όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά λογικό χρονικό διάστημα, σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση της εθνικής άδειας, ε, άρθρο 25, παράγραφος 5, Θεωρώ ότι για να υπάρξει πραγματική εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν επιθεμητό να προβλέψουμε στον κανονισμό ένα ε, μοναδικό αριθμό αδειών που θα δίνονται από όλα τα κράτη-μέλη και που ε, να έχονται στην αμοιβαία αναγνώριση του προϊόντος. Ό,τι αφορά τις ετικέτες, δεν θεωρώ ότι ο αριθμός ε, των αδειών όλων των βιοκτώνων που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αναφέρεται στις ετικέτες. Πρόκειται για μια πληροφορία που δεν έχει κανένα νόημα για την ασφάλεια του καταναλωτή. Αν ε, όμως ε, ένας ε, επιλέξει, κάποιος επιλέξει διαφορετικό προμηθευτή θα πρέπει να αλλάξει και ετικέτα γιατί αλλάζει το νούμερο της άδειας της ουσίας που έχει εγκριθεί σε ό,τι αφορά το παράλληλο εμπόριο θα έπρεπε να περιοριστεί σε προϊόντα που έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνουν τις ίδιες δραστικές ουσίες. Εγώ λοιπόν ε, δεν ε, είμαι σύμφωνος με την πρόταση της Κομισιόν. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα έπρεπε να εισαχθούν και στοιχεία που αφορούν την προστασία και την ανταλλαγή των δεδομένων για να αποφύγουμε το φαινόμενο του free riding και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ανακτήσουν τις επενδύσεις ε, που έχουν κάνει για την ανοδιότηση και την καταγραφή των βιοκτώνων και των δραστικών ουσιών. Σε σχέση με την εμπιστευτικότητα των ε, πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ε, διοδότηση, άρθρο 55 παράγραφος 2, θεωρώ ότι στο κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να είναι απόρριτες, πρέπει να προσθεθούν και η ημερομηνία της έκδοσης μιας άδειας και η ημερομηνία λήξης της. Το να διαδίδονται πληροφορίες για τη διάρκεια της αδειοδότησης ε, είναι ευαίσθητα εμπορικά πληροφορία κατά την ε, δική μου άποψη και θα πρέπει να διατηρείται απόρριτη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτόρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη, καθυστέρησα λίγο να έλθω. Εγώ θέλω να παρέμβω για το θέμα αυτό, γιατί είμαι εισηγήτρια στην ΕΝΚΟ για τον κανονισμό αυτό. Έτσι λοιπόν ε, χαίρομαι που στην έκθεση του κυρίου Καρίν βλέπω να έχουμε ένα καλό σχέδιο γνωμοδότησης με το οποίο συμφωνώ. Σύμφωνα με τη θέση που υποστηρίξαμε στην ΕΙΜΚΟ ε, αυτό εδώ το σχέδιο με βρίσκει σύμφωνο, αν και συζητήσαμε και άλλα επιχειρήματα. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του προ την έρευνα που πρέπει να απλουστευτεί και να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και συμφωνώ με την αναγκαιότητα να διευρύνουμε τη διαδικασία, ε, την κεντρική διαδικασία διοδότησης. Όμως πρέπει να εργαστούμε επί του κριτηρίου που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καταλήξουμε σε αυτή την επιλογή. Η λύση που προτείνεται από τον Σεγητή για μένα είναι αποδεκτή. Όμως υπάρχουν και άλλες προτάσεις ε, και από την πλευρά των κρατών μελών που τις λαμβάνουμε υπόψη, τις εξετάζουμε. Ίσως θα έπρεπε να αξιολογήσουμε και την καταλληλότητα μιας μελέτης που να μελετά το πιθανό αντίκτυπο της διεύρυνσης της κοινωτικής διαδικασίας επί της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και επί του περιβάλλοντος. Αυτό θα μας επέτρεπε να επιλέξουμε την καλύτερη μέθοδο. Είναι σημαντικό όμως για μένα να διατηρήσουμε τη δυνατότητα επιλογής μέσω της εθνικής αδειοδότησης ή της κοινοτικής αδειοδότησης για να μην δημιουργήσουμε μειονεκτήματα για ορισμένους πρωταγωνιστές. Πάντως ε, θεωρώ ότι για το μέσο συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να προβλέψουμε τη χρησιμοποίηση χρήση αφού θα έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία με τη χρήση ενός προϊόντος και για να μην δημιουργήσουμε υπερβολικά απαγορευτικούς όρους για όσους ε, σήμερα ε, μπορεί να χρειαστούν και πάνω από πέντε χρόνια για την καταγραφή ενός προϊόντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κομισιόν θέλει κάτι από αυτού, ο κύριος Πάλτ. Σύντομα παρακαλώ. Μάλιστα, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε καλωσορίζουμε την, το σχέδιο έκθεση ε, του εισηγητή που περιλαμβάνει διάφορα χρήσιμα στοιχεία και ευκρινήσεις. Ιδίω όσον αφορά τις ε, ε, τροπολογίες για τις παραλλαγές, ε, που φαίνονται σημαντικέ, καθώ επίση για την έρευνα και την ανάπτυξη και διάφορε από τι διαδικασίε και τι προθεσμίε. Δύο προβλήματα έχουμε. Το ένα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσίες που έχουν βέβαια μια εσωτερική δομή και θα πρέπει να γίνει σεβαστή όταν του ζητούμε κάτι. Και επίσης οι τροπολογίες 21 και 23 που αφορά τις προθεσμίες για την Κομισιόν για την Επιτροπολογία που μου φαίνεται ότι δεν είναι συμβατή με υποχρεώσει που έχουμε να έρθουμε σε επαφή και με εσά και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ και ιδίω γιατί ήσασταν τόσο σύντομο. Ο ζητητή μου θέλει να δευτερολογήσει, παρακαλώ. Μάλιστα, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, διατύπωση έκθεσης, είτε διότι ήρθαν σε άμεση επαφή με, τη, με μένα, είτε γιατί παρουσίασαν εδώ τις απόψεις τους. Από όλες τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής, έχω δημιουργήσει την εντύπωση ότι η συνάδελφοι είναι πάρα πολύ θετικοί όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθώ. Πράγμα που μου αποδεικνύει την επιδοσή τους στο έργο που πραγματοποιώ. Αν εξάζω πολύ γρήγορα τα θέματα που παρουσιάστηκαν, έχω να πω ότι υπάρχονται στις κατηγορίες ορισμού ε, τελεί τέλη, στοιχεία, δεδομένα. Αυτά είναι λίγο πολύ νομίζω τα θέματα που έθιξαν όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στη συζήτηση. Τα περισσότερα τα θέματα που εθίγησαν ανεμετωπίζονται από τις τροπολογίες που έχουν προσαρτηθεί στην γραμμοδότηση. Βέβαια, είμαι ο μόνος που θα παραδεχτώ ότι οπωσδήποτε ε, οι τροπολογίες μπορούν να βελτιωθούν. Και όσοι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες, θα χαρώ πάρα πολύ να τις δω γιατί ίσως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για κάποια σημεία. Όπως είπα όμως και εισαγωγικά, τα περισσότερα θέματα που εθίγησαν αντιμετωπίζονται με στροπολογίες που έχω υποβάλει. Τούτου λεχθέντος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στην προσέγγιση που θέλει να ακολουθεί οι συνάδελφοι. και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν αυτόν τον τόσο επικοδομητικό διάλογο με μένα μέσω και του γραμματεία μου και θα καταλήξουμε σε μία θέση που θα ικανοποιεί όχι όλους, αλλά τους περισσότερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο τη ημέρα τη διάταξη, χρηματοδοτική συνδρομή γνώση για την παραπλησμό των μονάδων 1 4 του πυρηνικού σταθμού Κοσλοντούι στη Βουλγαρία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά 10 λεπτά το χρόνο μας. Δεν είναι τόσο τραγικό ακόμα, αλλά αν το κάνουμε κάθε φορά θα έχουμε προβλήματα. Δεν σχετίζεται με την έκθεση αυτή, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να μην μακρηγορούμε ιδιαίτερα. Κυρία Χάμς έχει το λόγο, πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την έκθεσή μου πολύ σύντομα. Καταρχήν να σας πω περί τι πρόκειται. Έχουμε κάνει μια πρόταση για έναν κανονισμό και με τον κανονισμό αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, περαιτέρω ροή οικονομικής βοήθειας για, την, ε, για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού στο Κοσλοντούι στη Βουλγαρία. Θα σας πω ποια είναι τα βασικά σημεία. Αυτή η οικονομική ροή θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Ως ε, ε, εισηγήτρια το αναφέρω αυτό στην εκθεσή μου, αλλά θα ήθελα στον κανονισμό αυτό να ξεκαθαρίσουμε πώς έχει ε, εξελιχθεί η χρήση των κονδυλίων μέχρι τώρα και προς ποιο βασικό σκοπό απεστάλησαν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μιλούμε για την ασφάλεια των Βουλγάρων πολιτών και πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως προς αυτό λοιπόν, έχω αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί μέσω αυτού του κανονισμού. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Έχω αποστείλει έναν κατάλογο με τι ερωτήσει αυτέ στην Κομισιόν. Χτες ήρθα σε επαφή με συνεργάτες από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να, να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Σήμερα το πρωί έκανα μια πρώτη επαφή με τους ε, σκιώδεις συγητές. Η κυρία Σαποντιέ είναι... Ε, ήταν πολύ γρήγορη και οι, οι, οι ε, εξεκολουθούν να προωθούν την ε, εργασία, συμφώνησαν με αυτά που έχω υποβάλει εγώ στην έκθεσή μου. Θα είναι λοιπόν ε, μια έκθεση η οποία θα πάει αρχές Φεβρουαρίου στην, ε, στις μεταφραστικές υπηρεσίες και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερα κανθόδες θέμα το οποίο θα προκύψει. Το μόνο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικέ εκθέσεις για την ε, στρατηγική ε, παροπλισμού από τη Βουλγαρία, ε, τη χρηματοδότηση, την νέα χρηματοδότηση, θα πρέπει να την, να, να ξαναδούμε, να την ξαναμελετήσουμε πιο προσεκτικά. βασικό σημείο στην έκθεση βέβαια είναι να συμφωνήσουμε ως προς αυτό και να δούμε γιατί πώς μάλλον θα κινηθούν τα χρήματα, τα κονδύλια για, την, ε, για τον παροπλισμό των ε, μονάδων και γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να αποστέλουμε τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλφίν έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάρμς που μας ε, παρουσίασε τις απόψεις της για το θέμα. Θα ήθελα να βασιστώ σε μια προσέγγιση έναντι της απόφασης της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια επιπρόσθετη αντιστάθμιση για τη Βουλγαρία καταρχήν θα έπρεπε να είναι στο ύψος ε, της ενίσχυσης για τον παραπλησμό, όπως δόθηκε σε άλλες χώρες, Λιφανία και Σλοβακία, και θα έπρεπε να συνεχιστεί μετά το 2009. Τα μέσα τα κονδύλια αυτά θα έπρεπε από τις αρχές ε, να διοχετευτούν σε ένα ειδικό ταμείο όπως ε, έγινε με τις άλλες χώρες και θα χορηγηθούν τα κονδύλια για συγκεκριμένε δράσεις για τον παροπλισμό. Και άλλα κονδύλια θα εκπονηθούν, συγγνώμη, θα διοχετευτούν στην ε, δημιουργία πράσινων τεχνολογιών. Θα ήθελα να υποστηρίξω τα όσα είπε η κυρία Χάρμς. Δηλαδή, στο ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει πλήρη πληροφόρηση για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Η κυρία Χάνς λοιπόν θέτει το πρόβλημα με ιδιαίτερη σαφήνεια έτσι όπως εφαρμόζει και ίσως θα έπρεπε να απευθυνθούμε στην βουλγαρική κυβέρνηση για να μας δώσει συμπληρωματικά σχόλια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, τα νέα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακόμα ε, πυρηνικού σταθμού πρώτη γενιά και πρέπει να, τα, να τους παροπλήσουν. Και εμείς, όπως και η Βουλγαρία, έπρεπε να λάβουμε μια σημαντική, σοβαρή απόφαση για, την, για τον παροπλισμό αυτό έγινε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Ε, βέβαια αυτό οδήγησε και σε ανεργία, σε κοινωνικές εντάσεις και σε μια γενική ανησυχία, από απομόνωση μιας ολόκληρης περιφέρειας. Γι' αυτό αυτή η οικονομική ενίσχυση είναι πάντα απαραίτητη. Όπως το βλέπω εγώ, είναι αναγκαία σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών έτσι ώστε να εφαρμοστεί έγκαιρα το πρόγραμμα αυτό παροπλισμού, πρώτον αυτό, και δεύτερο, με τη βοήθεια αυτή την οικονομική, θα μπορέσει κανείς να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ του να μεταφερθούν σε άλλους τομείς αυτοί που εργάζονται τώρα στον πυρηνικό σταθμό. Οπότε θα ήθελα να πω ότι στην Κομισιόν ότι είναι πολύ καλό που ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και ευχαριστώ και την, την για, για το πόσο σημασία δίνει στο σημείο αυτό στην έκθεσή της. Γι' αυτό υποστηρίζω περαιτέρω την οικονομική ενίσχυση της Βουλγαρίας και το και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίσει αυτό, να συνεχίσει η ζωή των ε, κονδυλίων στην ε, χώρα αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρο. ιστορία ρεζουλτήρα εδώ Εδώ Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα μακρόν και τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν με τον παροπλισμό των τεσσάρων αντιδραστήρων στο Κοσολντούι στη Βουλγαρία. Έχουμε τεράστια ποσά ε, δηλαδή σε, έχουμε εκατομμύρια ευρώ άμεσων απελειών ε, λόγω του παροπλισμού. Η χρηματοδότηση ε, για τον παροπλισμό σταμάτησε και η Βουλγαρία δεν ήταν σε θέση να επιλύσει από μόνη της το πρόβλημα αλλά έπρεπε να λάβει τεχνική και χρηματοοικονομική βοήθεια. Αυτή η ε, οικονομική ενίσχυση είχε δοθεί στη Βουλγαρία μέχρι το 2009. Βέβαια, ίσως στις ε, μελλοντικές μας συζητήσεις να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί επιλέχθηκε το 2009 ως όριο. Πάντως ε, το ποσό ήταν ε, κατώτερο από τα κονδύλια που χορηγήθηκαν στα άλλα δύο κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το νέο αίτημα οικονομικής αρρωγής ε, ίσως θα μας θέσει σε ισότιμη θέση με τα άλλα δύο κράτη θα υπάρξει έκφραση της Ευρωπαϊκής Ελληνικής και θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που είναι ευρωπαϊκού βεληνικούς. Καθώς ε, συζητάμε τώρα το θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την έκθεση της κυρίας Χάρμς μας. Ε, είναι απαραίτητη η στήριξη αυτή αμέσως. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου να σα πω ότι συμφωνώ με τη θέση της κυρίας Χάνους και νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί της. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χέρτσοκ. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να επενθυμίσω την ιστορία του θέματος αυτού. Όταν ε, ε, συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουμε πρόσθετα κονδύλια στις χώρες αυτές ε, γιατί ο κ. Ε, Γιάνν Χούντατ από τη Σλοβακία και εγώ ως συγγήτρια είχαμε πει και νομίζουμε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο ότι το να κλείσουν αυτά τα εργοστάσια πριν να ιδρυθεί το Ταμείο του Περοπλισμού ε, έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να ιδρύσουμε αυτό το ταμείο, ούτε μπορεί να ε, ε, μπορούν να τιμωρηθούν οι Βούλγαροι, οι Λιθουανοί, οι Σλοβακοί, οι Σλοβάκοι, με συγχωρείτε, να τιμωρηθούν για το λόγο αυτό. Και χώρες ε, αυτές ε, τελικά πρέπει να φροντίσουν ε, να ρυθμίσουν αυτό το θέμα και τελικά η Επιτροπή αυτή αλλά και το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να λάβει την υποστήριξη από όλα τα μέρη. Εγώ εργάστηκα τα μάλα για το θέμα αυτό συμφωνώ με την προσέγγιση που ακολουθείτε εδώ και πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο ενωμένοι γιατί τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης τα ίδια τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκονται σε δινή θέση και πρέπει να βρούμε τα μέσα για να υποστηρίξουμε αυτές τις τρεις χώρες, τώρα τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι αυτά διακυβεύονται. Χαίρομαι που η Επιτροπή υιοθετεί μια τέτοια στάση υπεύθυνη και ελπίζω να μας βοηθήσετε στην Επιτροπή Προπολογισμού για να βρούμε τα κατάλληλα κονδύλια. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στην ε, Κομισιόν να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η πρότασή μας για αυτόν τον νέο κανονισμό έχει υποβληθεί, την έχετε, για διάφορους λόγους. Η χρηματοδότηση για τη Βουλγαρία για τον, αποκλει... τον ε, παροπλισμό των μονάδων στο Κοσλοντούι σταμάτησε πέρσι στην Ιγναλίνα και στον Μπορούνιτσε η χρηματοδότηση για τον παροπλισμό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2013 και θέλουμε με την πρότασή μας οι τρεις χώρες που πρέπει να απολαμβάνουν τις αλληλεγγύες μας να βρεθούν σε ίση θέση με τις υπόλοιπες για το χρονικό αυτό λοιπόν διάστημα έχουμε προτείνει 300 εκατομμύρια ευρώ για τον παροπλισμό. Γνωρίζετε τα προγράμματα, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Χάρμς αν υπάρχει ανάγκη για διευκρινήσεις ό,τι αφορά τη βουλγαρική πλευρά, τότε θα πρέπει όντως αυτό να το τονίσουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι οι βουλγαροί α, συνομιλητές μας θα μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες που ζητούμε στις ε, συνθήκες ε, ένταξης ε, αναφέρεται σαφώς ότι ο παροπλισμός θα πρέπει να συμπληρωθεί και για διάφορους λόγους και για το Κοσλοτούι πρέπει να πω ότι για παράδειγμα με, το, με το κλείσιμο αυτό των, των βασικών ομα, μονάδων 1 ως 4 θα αλλάξει και θα υπάρξουν ε, ή πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επενδύσεις. Απ' την άλλη, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με το Λονδίνο και, τους, ε, και τον χρηματοδότη από το Λονδίνο που δίνει τα, μέσω ημών τα χρήματα, θα καταλάβουν ότι η ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά προγράμματα, ειδικά για τη Βουλγαρία, είναι τα βασικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται στους υπόλοιπους εταίρους. Σύντομα, για να μην ε, σπαταλώ το χρόνο σας, υποστηρίζουμε και Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την γενική προσέγγιση και, τις, ε, και, τον, ε, και, τους, και τους στόχους που έχουμε θέσει. Θέλουμε την υποστήριξή σας και έχουμε υπόψη μας να μην γίνει προαίρεση η ασφάλεια. Πρέπει να, είναι ε, πρέπει να την εγγυηθούμε και βεβαίως να υπάρξει σαφής και απρόσκοπτος παροπλισμός των μονάδων στο Κοσλοντούι και να ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξη που λάβαμε για την, ε, την προηγούμενη χρονιά, για την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια, η οποία τώρα θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Ε, περιμένουμε την πρώτη, το πρώτο σχέδιο έκθεσης και με αυτά που αναφέρει η κυρία Χαρμ στην έκθεσή της, είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί αισίως η διαδικασία αυτή. Αυτή είναι η τελευταία μου φράση πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από το Συμβούλιο. Ελπίζουμε πριν, να γίνει, πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα να γίνει αυτό. Οπότε το Μάιο να μπορέσουμε να καταλήξουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο, να μπορέσετε μάλλον εσείς να καταλήξετε στο Κοινοβούλιο σε μια απόφαση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς αν θέλει και πάλι το λόγο. Για να δώσω ένα παράδειγμα γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα για το αν δηλαδή υπάρχουν ε, αρκετά χρήματα από αυτά που, ε, που ε, δίνονται για τον παροπλισμό. Στις μονάδες 3 και 4 στο Κοσλοντούι έχουν μεταφερθεί αρκετά τμήματα του ε, σταθμού έχουν ε, αποφορτωθεί ε, και βρίσκονται προς διάθεση εκεί επί τόπου στο Κοσλοντούι. Αλλά δεν υπάρχει εντωμεταξύ ενδιάμεση δυνατότητα αποθήκευσης. Αυτή θα πρέπει να υπάρξει, να δημιουργηθεί από την αρχή. Αυτό είναι κάτι όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι έτσι μόνο θα εξασφαλίσουμε σαφή και σίγουρο παροπλισμό μέσω αυτής της οικονομικής ενίσχυσης. Να μην υπάρξει δηλαδή υποχρηματοδότηση, αλλά επαρκής χρηματοδότηση. Κατά τα λοιπά, αυτή η συζήτηση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τώρα τις λεπτομέρειες που θα προκύψουν θα τις ε, περιμένω με χαρά πρέπει για το Κοσλοντούι να προετοιμαστούμε καλά για την διαδικασία αυτή παροπλισμού, γιατί υπάρχει και η σχετική οδηγία η οποία θα υποβληθεί από την Κομισιόν το Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχουν και πρότυπα ασφάλειας, τα οποία ανέφερε η Κομισιόν για, τον, για τους πυρηνικούς σταθμούς. Αυτά τα πρότυπα δεν βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Και νομίζω ότι αυτό έγινε σαφές και από την ε, ε, ακρόση που κάναμε τον κύριο Ότιγκερ. Αυτός θα είναι ο στόχος μας για τον επόμενο χρόνο, να φροντίσουμε να υπάρχουν υψηλά πρότυπα. Είμαι πάντως πολύ ικανοποιημένοι με το πώς έχουμε ξεκινήσει να διαχειριζόμαστε το θέμα αυτό του Κοσλοντούι και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ροή των πληροφοριών που μας έχει δώσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έκλεισε λοιπόν και το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Πάμε στο σημείο 13 και 14. Θα τα δούμε από κοινού ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, τροποποίηση τη οδηγία και του κανονισμού. Ο κύριος Χαρτζημαρκάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ αντικρουόμενο θέμα και πολιτικό καυτό. Εγώ ήμουν μέλος ε, του Φαρμακευτικού Φόρου, Φόρουμ και παρακολούθησα τις εργασίες για τρία χρόνια. Γενικώ πώς η πληροφόρηση των ασθενών είναι ένα παλαιό θέμα. Ήδη ξεκίνησε η συζήτησή του από το 2003 στο Κοινοβούλιο. Ε, κατέρευσαν οι συζητήσεις τότε και ελπίζω αυτή τη φορά να μην καταρρεύσουν. Θυμόμαστε όλοι την ακρόαση με τον Επίτροπο Νταλή στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Εκεί δεν, έχει, δεν είχε υπάρξει καμία σαφής απάντηση για το αν θέλει να αποσύρει την πρόταση ή όχι και δεν υπάρχει κανένα λόγο να την αποσύρει. Όλοι ξέρουμε ότι το πακέτο για τα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλα σημεία αποτελείται από, τρία, από τρεις τομείς. Ε, τα δύο είναι, τα δύο είναι ok, ε, δεν έχει υπάρχει πρόβλημα. Αυτό όμως είναι λίγο προβληματικό, γιατί αυτό είναι αυτό που αφορά και ενδιαφέρει τους ασθενείς. Να μπορούμε δηλαδή να δίδουμε ε, τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες για αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, για την υγεία τους, για τα φάρμακα που λαμβάνουν. Και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην ε, πολιτική πληροφόρηση του γιατρού. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους γιατρούς στην Ευρώπη. Μόνο 15 λεπτά χρόνο έχουν οι γιατροί της Ευρώπης κατά μέσο όρο για να ασχοληθούν με τους ε, ασθενείς τους. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ λίγο και πρέπει να ενισχύσουμε την πληροφόρηση που δίνεται έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να, να γιατρευτεί από την ασθένεια που τον ταλαιπωρεί. Γι' αυτό την, ε, έχει κάποια ε, καλά σημεία η πρόταση. Πρέπει λοιπόν να τη συμπληρώσουμε και με όσα λείπουν. Να... Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις οι οποίες αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα και παρεκκλίνουν πολύ από όσα εγγυόμεθα εδώ στο κείμενο. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει σαφής πολιτική από τις, ε, από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τον ασθενή. Γιατί το θέμα αυτό της πληροφόρησης των ασθενών είναι πάρα πολύ περίπλοκο και πάντα βρίσκεται υπό την προαίρεση ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί είναι διαφήμιση. Δεν μπορούμε να το δώσουμε ως πληροφορία αυτό. Πολλοί στην ε, συνάδελφη στο φαρμακευτικό φόρουμ, το λέει και η έκθεση, έχουν ε, πραγματικά ασχοληθεί με αυτό και υπάρχουν, ε, υπάρχουν πληροφορίες που δεν είναι διαφημιστικές. Μιλούμε για ουδέτερες, αξιόπιστες, αντικειμενικές πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες, Έχουμε και έναν έλεγχο εξάντε ο οποίος προβλέπεται και καμία πληροφορία για ένα φάρμακο για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή δεν μπορεί να δίνεται χωρίς επαρκή έλεγχο ή έγκριση από, τους, από τις αρχές. Η έκθεση το λέει και η πρόταση το λέει, η αρχή αυτή ορίζεται από το κράτο μέλος. Το κράτο μέλος το κράτος μέλος είναι ελεύθερο να ορίσει την αρχή. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένας ένα ενδιάμεσο ε, σταθμός. Δηλαδή η αρχή ε, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ε, πληροφορίες, να τις ελέγχει και να τις εγκρίνει ή όχι. Το βασικό λοιπόν σημείο εδώ παραμένει το, ε, το φύλλο οδηγιών. Ποιο διαβάζει από εσά τα φύλλα οδηγιών στα φάρμακα που παίρνετε με, την ο, με τη συνταγή. Ο Παουλ Ρούμπικ σήκωσε το χέρι του, αλλά μάλλον είναι ο μόνο που το κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι, και εγώ επίση, δεν το διαβάζουμε με ευχαρίστηση γιατί φοβόμαστε από αυτά που διαβάζουμε για πολλού, το φύλλο οδηγιών ε, είναι ένα έγγραφο που είναι γραμμένο από νομικού για νομικού. Δεν είναι κατανοητό, δεν είναι σαφέ. Και προ το παρόν, με τι πληροφορίε και την πολιτική πληροφόρηση για του ασθενεί, για του πολίτε, δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι τα ε, φύλλα οδηγιών. Πρέπει να, πρέπει να αλλάξουν. Δεν μιλούμε για διαφήμιση. Μιλούμε για το πώ μπορούμε να διευρύνουμε τι πληροφορίε που περιλαμβάνει το φύλλο οδηγιών, πώ θα γίνει αυτό μέσω μια κεντρική αρχή, πώ μπορούμε να ενισχύσουμε με ίσω κάποια γραφικά ή να τα εξυγχρονίσουμε τα φύλλα γιατί υπάρχει τεχνολογία στην Ευρώπη και αυτό είναι θέμα ιστορική αγορά. Σε διάφορε χώρε υπάρχουν άλλε δυνατότητε να συμπληρωθούν τα φύλλα Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μια ενοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών και θέλουμε τα φιλοδιό να βρίσκονται και online, στο ίντερνετ. Έτσι ώστε ο καθένα να μπορεί στη γλώσσα του να έχει πρόσβαση να διαβάζει αυτά τα οδηγιών, τα καινούργια. Ας πούμε για κάποια σκευάσματα για αναπνευστικά προβλήματα, να ξέρει κανείς πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει σωστά το σκεύασμα αυτό, τη συσκευή. Μιλούμε δηλαδή για τη σωστή χρήση και μιλούμε και για την αποτελεσματικότητα του ασθενούς. Έχουμε 400 ε, ε, εγκεκριμένα φάρμακα. Μιλούμε για ε, αρχές οι οποίες θα συμπληρώσουν τα, και θα, που εγκρίνουν και συμπληρώνουν τα φύλλα οδηγιών και επίσης ως συμβαστική πρόταση θα ήθελα ήδη να πω ότι αυτό το ακαθόδες θέμα της, των δημοσιεύσεων σχετικά με την υγεία, δηλαδή έντυπα, τα οποία ξεπερνούν τα όσα αναφέρονται στις, στα φύλλα οδηγιών, θα μπορούσαμε να τα δούμε μεταγενέστερα. Γιατί ε, αυτό είναι το ακαθόδε θέμα. Υπάρχει εδώ η κατηγορία ότι μέσω αυτών των ε, ε, δημοσιεύσεων υπάρχει κρυμμένη διαφήμιση. Αν συνέβαινε αυτό, τότε μπορούμε να το διαγράψουμε, εννοείται. Και κάτι τελευταίο, ανταλλαγή επιστολών μεταξύ φαρμακευτικών βιομηχανιών και ασθενού. Αυτό είναι ακαθόδε θέμα. Μπορεί η φαρμακοβιομηχανία να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα του ασθενού. Μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Αποκλείεται στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να γίνεται, αλλά μέσω μιας ενδιάμεσης ε, αρχής. Ε, γιατί, και βεβαίω θα χαρούν πολλοί αρχέ γιατί θα έχουν περισσότερη δουλειά, αλλά τουλάχιστον αποκλείουμε την, την άμεση επαφή φαρμακοβιομηχανίας ασθενού και έχουμε την δυνατότητα να πληροφορεί το ασθενή όταν έχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα να το αποστέλει στην αρχή η αρχή στη φαρμακοβιομηχανία και να λαμβάνει την απάντηση. Δηλαδή έχει το δικαίωμα ο ασθενή να, λαμβάνει τις πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε με στόχο τον, α, τον ασθενή, γιατί μιλούμε για δικαιώματα των πολιτών. Και εδώ θα πρέπει να, ήδη στον επόμενο γύρο να προχωρήσουμε με μια νέα συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή γιατί αφορά τους πολίτες της Ευρώπης. Μιλούμε για πρόσβαση σε πληροφορίες και την πρόταση αυτή, την πρόσβαση πρέπει να την εγγυηθούμε και βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε την διαφήμιση. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση. Υπάρχει ένα γεγονός. Η ΥΠΟΗ θεωρεί πως περίπου 50% των Ευρωπαίων ασθενών δεν γνωρίζουν σαφώς για το ποια, φάρμακα παίρνουν. Δεν το ξέρουν, ε, δεν γνωρίζουν τα φάρμακα. Οπότε πραγματικά πρέπει να αποφύγουμε ένα, μια, μια ασθενοπό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε την πρόταση αυτή με τροπολογίες. Αυτές οι τροπολογίες προσπαθούν, έχουν ως στόχο να καταδείξουν που είναι τα προβλήματα. Τροπολογία 20 εδώ μιλούμε για το ότι μπορεί να υπάρξει ε, προσφυγή έναντι των ε, αρνητικών αποφάσεων από τις ε, αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, τι μηχανισμός είναι αυτός. Πριν μιλούσαμε για κυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η προσφυγή μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου μπορεί να διαρκέσει δύο ή τρία χρόνια να ληφθεί μια απόφαση, μια νομικώ δεσμευτική πρόταση, παρόλο που οι κυρώσει μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κορέρα Δακάμπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι προτάσει του εισηγητή γενικά είναι καλές και οδεύουν προς την διακδέθυνση με τις δικές μας απόψεις. Γενικά είμαστε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής έτσι ώστε να αποφευκτεί η διάδοση ε, της διαφήμισης και να υπάρχει σύγχυση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Όμως υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις ακόμα. Είμαστε υπέρ της τροπολογίας 3 για την ενημέρωση του κοινού φυσικά, αλλά ε, διαφωνούμε για το να μπορούν να, να ανατεθούν υπεργολαβικά ε, οι αρμοδιότητες ενημέρωσης των ε, ασθενών από τις φαρμακοβιομηχανίες. Επίσης ε, επιτρέπεται να απαντήσει με ηχογράφηση η αρμόδια φαρμακοβιομηχανία στους ε, ασθενείς. Όμως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε δυσκολίες σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση. Γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τόσο εύκολα αυτό το είδος της απάντησης όπως τη γραπτή απάντηση. Επίσης επιτρέπεται να δίνονται πληροφορίες μέσω βίντεο. Ε, το βίντεο επιτρέπει με πολύ μεγάλη ευκολία να ε, διαβιβάζονται μηνύματα διαφημιστικού χαρακτήρα όμως ε, εδώ και πάλι θα μπλέξουμε το θέμα της ενημέρωσης με τη διαφήμιση. Έχουμε και άλλες ε, μικρές αποκλήσεις. Συμφωνούμε με τη γενική κατεύθυνση της πρότασης, αλλά θέλουμε να εγγυθούμε καλύτερη διάκριση μεταξύ της ενημέρωσης και της διαφήμισης, καλύτερο ορισμού των, επιτε... επιτετραμένων διάβλων και επίσης ε, δεν ε, θέλουμε να υπάρχουν ενδιάμεση για τη διάδοση των πληροφοριών. Δεν ξέρω, πρέπει να περάσω και στον κανονισμό. Πρόεδρε, είπατε ότι θα τα δούμε από κοινά τα δύο αυτά θέματα. Μπορώ να συνεχίσω, ωραία. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Οι προτάσει του εισηγητή γενικά είναι καλέ και οδεύουν προ την ίδια με αυτά που πιστεύουμε και εμεί. Προτείνει ο εισηγητή ε, να υπάρξει αύξηση ε, του κόστο ε, ε, του ΕΟΦ και αυτή η αναγκαιότητα χρηματοδότησης να αναλυφθεί μέσω του προπολογισμού της Ένωσης. Είναι ε, η διαδικασία αξιολόγησης να είναι πιο διαφανής ε, και να γίνεται με τρόπο και να καταπολεμούνται οι αντιφάσει. Και εδώ συμφωνούμε, όμω υπάρχουν κάποιε αποκλήσει. Προτείνει ο εισηγητή να μειωθεί η πρόθεσμη αξιολόγηση ε, από τι 60 στι 30 ημέρε. Εμεί αντίθετα προτείνουμε την αύξηση σε 120 ημέρε για να αποφύγουμε η έγκριση πληροφοριών εν γέννη να γίνεται σιωπηρά. Έτσι εγγυόμαστε την καλύτερη ενημέρωση, πιο αξιόπιστε πληροφορίε και δεν ε, διατίθεται και ο κίνδυνος ε, να υπάρξουν ε, διαφημίσεις αν δεν τοποθετηθεί εν ευθέτω χρόνο ο οργανισμός. Γενικά συμφωνούμε με τον συγγητή, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η διεύρυνση της βάσης δεδομένων του Ιούντραφαν θα λειτουργεί, για να λειτουργήσει ως βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε μία βάση δεδομένων η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και όλα τα φάρμακα που εγκρίνονται, αδειοδετούνται από τις εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι διαθέσιμε σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάσουμε μία τροπολογία για τις προτάσεις μας αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαστε σύντομοι. Ξέρετε ότι ο Επίτροπος Ντάλι έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει την πρόταση, οπότε θα επικεντρωθεί περισσότερο στους ασθενείς, έτσι ώστε να καλύψει και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Βέβαια, προ το παρόν τώρα είναι δύσκολο, θα καταλαβαίνετε, για μια ε, υπηρεσία να εκφραστεί επί τόσων πολλών τροπολογιών. Βεβαίω το καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο κύριος Χατζημαρκάκη και πάλι. Σύντομα, Πρόεδρε. Ο κύριος Νταλίοντο το είπε αυτό. Χαίρομαι που θέλει να λάβει υπόψη του αυτά που ζητά το Κοινοβούλιο. Έχουμε κι εμείς ευθύνη δεν θέλουμε να αποσυρθεί η πρόταση. Τώρα, για τα σχόλια που ακούστηκαν. Η ε, αντίθεση που έχει ο κύριος Μπάλσο με την, ε, με τροπολογία 20 έχει να κάνει με τον κανονισμό που ανέφερε και ο κύριος Κορέα Δεκάμπος. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση. Μέσα σε 30 μέρες θα πρέπει να υπάρξει απάντηση. Αλλά εγώ είμαι διατεθειμένος να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αν δηλαδή θα ήταν καλύτερε οι 120 ημέρε ή τέλο πάντων κάτι ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ε, προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να υπάρξει απάντηση ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσει. Για τα βίντεο. Και αυτά πρέπει να εξετάζονται μέσω των σχετικών αρμοδίων αρχών. Για να μην υπάρχει υποψία διαφήμιση. Αν υπάρχει υποψία διαφήμιση, απαγορεύονται. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφέ στην έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει το, εκ των προτέρων έλεγχο. Γενικώ χαίρομαι που υπήρξε, υπήρξε αρκετή υποστήριξη και βεβαίω ε, περιμένω και τι ε, τροπολογίε σα έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν ε, συμβιβασμοί και θα του βρούμε του συμβιβασμού, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο τη διάταξη. Στον Αλφα θέλει κάτι να πει, Κύριε Κουτιέρε. Θέλετε να μιλήσετε? Συγγνώμη, ήμουν σε τρεις ε, συνεδριάσεις ταυτόχρονα και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τώρα το λόγο για να μιλήσω για την εκθέση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι η διαβούλευση που έλαβε χώρα ήταν θεαματική. Νομίζω ότι είναι ένας ε, τρόπος ε, ε, μπορεί να μας βοηθήσει στο να πείσουμε τον πληθυσμό ότι εργαζόμαστε κοντά του. Αυτό είναι ένα θέμα επικοινωνίας, όμως είναι ένα θέμα που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω να βάλω, να παρουσιάσω συγγνώμη και κάποιες τροπολογίες. Εγώ νομίζω ότι με μεγάλη λογική έχει λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, όπως και στο θέμα της ενημέρωσης. Όμως εγώ θέλω να επιμείνω στο ότι υπάρχουν τρόποι που έχει κοινωνία και θα πρέπει να προωθήσουν τα κράτη για να αποφευχθεί η άμεση σχέση ε, ασθενών με τις επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου λόγου χάρη. Αυτό υπάρχει. Όμως ε, τα κράτη θα πρέπει να κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πετύχουν. Εμείς ε, στην Ισπανία έχουμε το 112 ε, που ε, είναι μια τηλεφωνική γραμμή και μπορεί κάποιος να ζητήσει συμβουλές από το γιατρό. Εμένα μου συνέβη πολλές φορές στην οικογένειά μου στις 5 η ώρα το πρωί να πάρει κάποιος τηλέφωνο και ένας καρδιοπαθής και να ρωτήσει «Α, έχω αυτό το πρόβλημα» και μου λέει αμέσω ο γιατρός ποιο φάρμακο πρέπει να πάρω. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβό και είναι δυνατό μέσω του τηλεφώνου είτε οι περιφέρειες είτε τα αρμόδια κράτη να δρομολογήσουν τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η διαβούλευση με τον γιατρό να είναι κάτι πολύ εύκολο γιατί άλλος τρόπος δεν λειτουργεί. Είναι κάτι φτηνό και μπορεί να υλοποιηθεί. Επίσης, θέλω να θέσω μια ερώτηση στους συναδέλφους. Ε, στη χώρα μου τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική κρίση και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη εισβολή ε, διαφημίσεων των φαρμακευτικών προϊόντων. <laughs> Απόλυτη εισβολή. Και τελικά λέει, διαβουλευτείτε, συμβουλευτείτε το γιατρό σα. Όμω βάζει ένα κύριο ή μια κυρία που θέλει να πάει στο θέατρο, ε, παραδείγματο χάρη, έρχεται η πεθερά, του δίνει το φάρμακο και σε πέντε λεπτά θεραπεύεται. Ή θέλει να πάει σε μια γιορτή και τελικά μπορεί να το κάνει γιατί θεραπεύεται θαυματουργά μόλι πάρει το φάρμακο. Και αυτό είναι διαφήμιση που υπάρχει. Και εγώ νομίζω ότι προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο να μα δώσει καθοδήγηση αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή τη οικονομική κρίση αυξήθηκαν πάρα πολύ οι διαφημίσεις. Γιατί εδώ μιλάμε για κάποια πράγματα, αλλά διαφορετική πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε το σημείο αυτό. Προθεσμία για τι τροπολογίε. 3 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Παρακαλούμε όποιος έχει τροπολογίες να τη στείλει ως τότε. 15-16, σημεία 15-16. Πάμε στην φάρμακο φάρμακοεπαγρύπνηση, ούτε καν να το πω δεν μπορώ. Δύσκολη λέξη, δύσκολη. Λοιπόν, θα την κάνουμε από κοινού τη συζήτηση για τα δύο αυτά σημεία. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στην εισηγήτρια. Η κυρία Ριβάζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Τι σημαίνει η φαρμακοεπαγρύπνηση. Παρακολουθούμε τις παρενέργειες ε, των ε, φαρμάκων και τώρα παρακολουθούμε τις παρενέργειες των εμβολίων ε, για τη γρήπη H1N1. Πρέπει να δούμε ε, ουσιαστικά ότι η οδηγία αυτή προέρχεται με προβλήματα που είχαμε όπως με το τηλεδομίδι και το διελιστήλι που προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα σε, στις γυναίκες και είχαμε και πολλές ε, ατροφές μελών για τις έγκυες γυναίκες που το ε, χρησιμοποιούσαν ως ηρεμιστικό. Έτσι λοιπόν, ε, κατόπιν αυτών υπήρξε η φαρμακοεπαγρύπνηση και ήταν πρωτοπόρος η Ευρώπη έτσι λοιπόν μας προτείνει η Κομισιόν μια επικαιροποίηση αυτής της οδηγίας. Υπάρχουν ήδη κάποια καλά στοιχεία αλλά πρέπει και κάποια να βελτιωθούν. Καταρχήν πρέπει να επαγρυπνούμε για τις άδειες που τίθεται στην αγορά πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί είτε μιλάμε για ε, τις κλινικές δοκιμές ανάτι που μας επιτρέπουν ε, να εντοπίσουμε ήδη τις παρενέργειες και όταν ζητάμε ε, άδειες ε, για υπόρους θέσεις στην αγορά θα πρέπει να έχουμε εξαίρεση της εξαίρεσης δηλαδή πρέπει να αιτιολογούμε τι θα επιφέρει το νέο φάρμακο σε σχέση με το φυστάμενο. Το δεύτερο ε, είναι το εξή. Όταν διανέμονται τα φάρμακα, πώς γίνεται η αναφορά των ανεπιθυμητών ενεργειών, των παρενεργειών. Ε, σίγουρα οι επαγγελματίε τη υγεία εμπλέκονται σε αυτό, αλλά η διαπίστωση των γιατρών είναι ότι δεν ε, συμπληρώνονται τα δελτία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταπόκριση από του ε, επαγγελματίε του κλάδου για τι παρενέργειε. Έγινε μια συνάντηση με του επαγγελματίε του κλάδου, των, τη Ενώση, του υπευθύνου τη φαρμακοεπεργρήμψη και τι μα λένε οι γιατροί. Είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία εργασία, έχει πάρα πολλά χαρτιά, είναι πολύ γραφειοκρατική ε, και θα πρέπει να το κάνουμε από την αρχή. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε, να εμπλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερο του ασθενεί. Όταν ο ασθενή ε, παίρνει το φάρμακό του και ε, του εκδηλωθούν παρενέργειε, θα πρέπει να ενημερώσει κατευθείαν τι περιφερειακέ και εθνικέ αρχέ και ταυτόχρονα να ε, οθήσει και το γιατρό να εμπλακεί στην κοινοποίηση. Όμως θα πρέπει να μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στις εθνικές αρχές. Και ε, από μία μελέτη προκύπτει ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες έτσι από αυτές που αναφέρουν οι γιατροί. Έχουμε πιο πλούσια αξιολόγηση ε, για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι λοιπόν προστακίθουμε τώρα προβλήματα σε επίπεδο εργαστηρίων. Ε, τι ζητάμε αυτά τα φαρμακευτικά εργαστήρια να μην αποφεύγουν τα εθνικά ή τα περιφερειακά κέντρα για να δώσουν κατευθείαν τις πληροφορίες στο Ultra Vigilance. Θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά αυτό γιατί διαφορετικά τα εθνικά και τα περιφερειακά κέντρα θα βρεθούν με έλλειψη δεδομένων και ε, επί της ουσίας ε, αυτά ε, είναι που συνδέονται λιγότερο σε σχέση με την παρασκευή των φαρμάκων. Εγώ θα ήθελα να εμπιστευόμαστε πραγματικά τους θεσμού μας και τους εθνικούς και περιφερειακούς αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή ε, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα εθνικά, να ενισχύσουμε τα εθνικά και περιφερειακά κέντρα είτε με χρηματοδότηση για τις χώρες που μπορούν, ε, εθνική χρηματοδότηση είτε μεικτή χρηματοδότηση. Αλλά προσοχή να μην έχουμε μόνο ιδιωτική χρηματοδότηση. Γιατί Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατά του να ε, καταβάλλεται ένας φόρος επί των φαρμάκων, όμως ε, προσοχή, ε, γιατί υπάρχουν... Ε, κάποιες φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες ε, χρηματοδοτούν αποκλειστικά τα κέντρα. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε την κοινοποίηση, αλλά ζητάμε να υπάρχει και διαφάνεια, έτσι ώστε οι εμπειρογνώμονες των μη να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Η Κομισιόν μας προτείνει μόνο εδώ να συμμετέχουν οι εθνικές αρχές, οι επαγγελματίε ε, του κλάδου. Εμείς θέλουμε άνοιγμα αναφέρεται και σε μια επιτροπή ενισχυμένη φάρμακο υπραχνήπηση. Τώρα, πώ λειτουργεί αυτό, Υπάρχει μια ομάδα εργασία, μια ομάδα εργασία που είναι όμω άτυπη. Η Κομισιόν προτείνει μια συμβουλευτική επιτροπή. Συμβουλευτική επιτροπή που να κάνει συστάσεις ε, εδώ εμείς προτείνουμε κάτι διαφορετικό, μια επιτροπή αξιολόγησης που να έχει και αρμοδιότητες. Ε, ε, αξιολόγησης λοιπόν ε, της φάρμακοεπεραγρήμησης σε σχέση με τα δεδομένα της Utravigilance και βάσει και των δεδομένων που έρχονται από τα κράτη. Πώς θα είναι, ποια θα είναι η σύσταση. Η Κομισιόν προτείνει να έχουμε 10 άτομα που θα διορίζονται από τα κράτη, συν 5 άτομα που θα διορίζονται από την Κομισιόν η ε, κυρία Μάκαβαν ε, που έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στην Επιτροπή ΕΝΒΗ προτείνει να υπάρχει ένα άτομο που να εκπροσωπείται 27 κράτη. Εγώ κάνω μια διαφορετική πρόταση, η οποία λειτουργεί πολύ καλά σε ορισμένε χώρε. Είναι να έχουμε δύο σώματα. Δηλαδή, αν ε, εδώ ε, μιλώ για την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία αυτού που θα συστήσουμε. Να υπάρχει ένα σώμα εκπροσώπων ε, από διάφορα κράτη, φυσικά θα είναι εμπειρογνώμων, δεν θα βάλουμε εκεί ανθρώπου που δεν ξέρουν τίποτα για τη φαρμακοεπιγρύπνηση, και να υπάρχει και ένα σώμα επαγγελματιών τη υγεία και ένα συνδεόμενο σώμα, δηλαδή μάλλον από ενώσει. Εκεί μπορεί να συμμετέχουν άτομα από τι ενώσει καταναλωτών ή από του ασθενεί κτλ. Και ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι ενώσει αυτέ γνωρίζουν περί και νομίζω ότι με αυτά τα τρία σώματα θα υπάρχει αξιοπιστία. Παρά να έχουμε κάθε φορά τον εκπρόσωπο από μια χώρα Ποιο, πώς θα διοριστεί, από ποιον, με ποια κριτήρια κτλ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αξιοπιστία με αυτά τα τρία σώματα. Τώρα, ε, μιλήσατε για το φυλάδιο οδηγιών ε, στα φάρμακα ή κομισιόν προτείνει μία σύνοψη. Τι θα βάλουμε σε σύνοψη. Αν ε, έχουμε μία σύνοψη για να μην βάλουμε τις περιενέργειες, λέμε ότι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στους ασθενείς αν βάλουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Όχι, εγώ προτιμώ να έχω τις ανεπιθύμητες ενέργειες ε, και να ξέρω ότι α, αν μου εκδηλωθεί αυτό το έλεγε στο φυλάδιο. Επομένως ε, δεν είναι κάτι που πρέπει να με ανησυχεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπεύθυνε τώρα. Αν ε, ο ασθενή έχει άλλε ερωτήσει, μπορεί να απευθυνθεί στο γιατρό του. Αλλά... Εμείς θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν πιο πλήρε εσόκληση στο φυλάδιο οδηγιών. Μπορεί βέβαια ε, το πλήρες φυλάδιο να είναι και στο διαδίκτυο και στο εσωτερικό του φαρμάκου να έχουμε ένα πιο συνοπτικό φυλάδιο. Αυτά λοιπόν για τη φαρμακοπαραγρύπνηση και θέλουμε να είναι κάτι αντιληπτό από όλου. Γιατί αν έχουμε καλή φαρμακοπεριγνώμηση, θα έχουμε και καλή ασφάλεια των ασθενών και οι ασθενεί θα εμπιστεύονται τα φάρμακα και τα εργαστήρια. Σα ευχαριστώ. Στον Χατζημαρκάκη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Πράγματι δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τι περισσότερε από τι παρατηρήσει τη εισηγητρία. Πράγματι, οι εθνικέ τράπεζε δεδομένων πρόκειται να καταργηθούν λίγο πολύ. De facto. Και από σκοπιά των ε, ασθενών θα πρέπει να υπάρχουν όμως κάποιες τράπεζες δεδομένων που θα είναι πιο ακριβείς και πιο ενήμερες και θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα προβλήματα αν υπάρχουν. Αναφέραμε εδώ στο άρθρο 107 τη οδηγία. Όσον αφορά τον κανονισμό, αξίζει πραγματικά να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύνου στα πλαίσια της φαρμακοϊπαχρύπνησης. Είναι κάτι που μπορούμε να το μελετήσουμε και να υποβληθεί και σχετική πρόταση. Όσον αφορά το άρθρο 21, Αναφέρεται στην προσωρινή χορήγηση της έγκρισης για την εμπορία. Αυτό θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο εάν υπάρχουν επιπτώσεις για τη μη τήρηση των ε, όρων που τίθενται. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή επιπτώσεις αν κάποιος δεν τηρεί αυτά που λέγονται. Και τώρα για το άρθρο 23 που αναφέρατε ποια ε, ε, φαρμακευτικά αντισυντάγματα θα πρέπει να ελέγχονται πιο έντονα. Εάν γίνεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να βάλουμε κάτι απάνω στο, στη συσκευασία για να φαίνεται αυτό ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στον ιατρικό τομέα και οι ασθενείς να το γνωρίζουν. Αυτές είναι κάποιες ε, προσθήκες που θα μπορέσουμε να τονώσουμε. Ευχαριστώ, συνέλφο Μπάλτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 3 και 5 όπου λέγεται ότι το 5% των στανών που εισάγονται στο νοσοκομείο εισάγονται λόγω επιπτώσεων από φάρμακα. Πολύ υποφέρουν από το τέτοιο. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι κάτι που το συζητήσουμε και στο παρελθόν και ήδη στο παρελθόν είχαμε πει ότι θα πρέπει ε, η φαρμακοεπαγρύπνηση να εξασφαλίζεται από πλευρά εμπειρογνωμόνων. Γιατί η φαρμακοβιομηχανία είναι δεύτερη μετά την οπλοβιομηχανία όσον αφορά τα κέρδη. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε και γι' αυτό θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια που εργάστηκε τόσο σκληρά θα μπορούσε να μου πει κατά πόσο και εκείνη πιστεύει ότι αυτέ, αυτοί οι εργασμοί είναι πραγματικά τόσο ανεξάρτητοι. Ευχαριστώ κορέα κάπως. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτά τα δύο νομοθετήματα είναι πολύ σημαντικά εμείς είμαστε θετικοί απέναντι στις προτάσεις της εισηγήτριας. Γενικά συνάδουν με τις ανησυχίες μας. Υπάρχουν κάποιες θετικές στοιχείες, όπως ε, να διαχωριστεί το τμήμα ε, των ουσιαστικών πληροφοριών στο φυλάδιο, γιατί αυτό μπερδεύει τον αναγνώστη και στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν δικέ του αρμοδιότητες για τη φαρμακοεπραγνύμπνηση να περιοριστεί ε, ουσιαστικά ε, το, ο τρόπος που δίνει απάντηση η βιομηχανία στους ασθενείς, ε, να ε, έχουμε όρους για την αδειοδότηση, αν δεν γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες και να βελτιώσουμε το μηχανισμό της πρόσβαση στα δεδομένα για τις παρενέργειες. Όμως έχουμε δύο σχόλια διαφορετικά. Καταρχήν για τους περιορισμούς ε, σε σχέση με τη θέση νέων φαρμάκων στην αγορά αν αυτά δεν παρουσιαστούν ως τα καλύτερα, την best in class. Ε, αυτό μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ε, γιατί μπορεί να αποτελέσουν κόλλημα στην καινοτομία και στον ανταγωνισμό και θα θέσουν μια μια πολύ μεγάλη έρηδα μεταξύ των κατόχων, ε, των παλιών κατόχων ε, της άδεια με τους νέους ε, ανταγωνιστές και θα δημιουργηθεί η ποικιλομορφία κριτηρίων μεταξύ των διαφορών κρατών μελών και επομένως θα ζημιώσει την απαραίτητη εναρμόνιση γιατί θα υπάρχουν κάποια κράτη που θα έχουν πιο φιλελεύθερη στάση στην εισαγωγή νεοφαρμάκων αλλά λιγότερο. Έτσι λοιπόν χάνουμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Έτσι λοιπόν εδώ μπορεί να υπάρξουν ε, αποκλήσει στο θέμα αυτό. Τώρα, το θέμα του reporting, ε, της ε, κοινοποίησης από τους κατόχους των αδειών ότι περνά στις ε, εθνικές αρχές ε, έναντι της Ευρωπαϊκής Αρχής. Αυτό ουσιαστικά αντίκειται στο μηχανισμό απλούστευσης προτείνεται από την Κομισιόν. Η Κομισιόν προτείνει απλώς να υπάρχει μια μεταφορά στο Udra Vigilance και ε, μάλιστα προτείνει να δίνονται και κίνητρα. Αυτά σε σχέση με την οδηγία τώρα για τον κανονισμό. Γενικά συμφωνούμε και πάλι. Θα ήθελα να τονίσω όμως ένα σημείο στο οποίο διαφωνούμε. Η συγγήτρια υπερασπίζει να υπάρχει αποκλειστικά δημοσιο σύστημα χρηματοδότησης, αλλά εμείς κατανοούμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο άχθος ε, για τους ε, εθνικούς και για τον ευρωπαϊκό οργανισμό και επίσης ε, θα αναλάβουν και πολύ μεγάλη ευθύνη οι κατόχοι των αδειών, η βιομηχανία δηλαδή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης που θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο. Το να επικεντρωθούμε τώρα εδώ στη δημόσια ευθύνη ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να αναλυφθούν όλες οι ευθύνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούμε ότι σε οικονομικό επίπεδο δεν θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση. Η κυρία Κουτιέρης, παρακαλώ. Υπάρχει και το θέμα της ε, φαρμακοεπαγρύπνησης που με ανησυχεί πολύ. Εγώ έχω παρουσιάσει κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει ε, να είναι στο μέσο, πρέπει να τονωθήσουμε θεματικά στην έρευνα για το... να υπάρχει ουσιαστικά εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων ε, ενεργειών. Ε, κοιτάξτε, αυτό το θέμα δεν μπορούμε στην πραγματική ζωή να το διαχωρίσουμε από τη φαρμακογρήγνηση, δηλαδή από την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η διάγνωση. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο και ακριβώς ε, στη σύνδεση που έχει με το αποτέλεσμα του φαρμάκου. Ξέρουμε, παραδείγματο χάρη, στην, σε εξετάσει του καρκίνου προκύπτουν πολλές, πολλά δικαρκίνου. Υπάρχουν πολλά δικαρκίνου, όμως πολλά νοσοκομεία δεν έχουν τόσο αναπτυγμένο σύστημα ε, έτσι κάνουν κάποιες διαγνώσεις που καλύπτουν ένα τομέα, αλλά δεν ε, μπορούν να κάνουν κάποια συγκεκριμένη διάγνωση με ακρίβεια. Αυτό εξαρτάται από το εργαστήριο που έχει το νοσοκομείο. Κάποιες ε, ομάδες γιατρών που εργάζονται, που ασχολούνται με το καρκίνο του στήθους, σε διεθνέ ε, επίπεδο ζητούν συνήθω δεύτερη διάγνωση για να δουν αν πράγματι χρήζει αυτή τη θεραπεία στο άτομο και πολλές φορές έχουν αποκλείσει ε, θεραπεία σε ορισμένα άτομα γιατί δεν είχε γίνει σωστά η διάγνωση. Δηλαδή, ακόμη και στον ασθενή ε, ο οποίος θα ε, δώσει ε, τελικά κάποια δεδομένα για τη φαρμακοπεγκρύπληση, δεν έχουμε τα στοιχεία του του έχει γίνει ορθή διάγνωση. Έτσι λοιπόν, εμένα μου φαίνεται ζωτικό για ορισμένα είδη ανάλυσης να απαιτούμε να γίνεται σωστή διάγνωση, όχι μόνο γιατί μπορεί να υπάρχει λάθος, αλλά γιατί μπορεί το χάρη κάποια άτομα να επιβληθεί κάποια σκληρή θεραπεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ε, σχετίσουμε τα κριτήρια της ποιότητας με έναν έλεγχο της καλύτερης διάγνωσης αν, ε, αν έχουμε επιλόγου χάρη ένα κατάλογο ατόμων ε, που πεθαίνουν επειδή υπάρχει κακή διάγνωση και έχουν πάρει λάθος φάρμακα, αυτό θα ήταν τρομερό. Κάθε φορά οι πελάτες γίνονται και όλο πιο επιθετικοί και μάλιστα έχουμε ε, και δικηγόρους οι οποίοι τελικά ζητούν να λογοδοτήσει το δημόσιο σύστημα. Όμως εγώ νομίζω ότι είναι θεμελιώδες αυτό το θέμα της διάγνωσης. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνάδελφος Ερτορία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να στεθώ σε ένα σημείο για τη φαρμακοπεραχλήπνηση με μια εισαγωγή. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι ε, όταν συζητούμε τα θέματα αυτά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μάλιστα όταν μιλάμε για ανθρώπους τόσο πολύ πιο προσεκτικοί είμαστε. Όταν ε, εμεί μιλάμε για φάρμακα, όχι μόνο ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του θέματος, αλλά μιλάμε και για ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι εκείνη τη στιγμή λόγω κάποιας νόσου. Έτσι, λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να συζητούμε τέτοια θέματα <laughs> με τον ίδιο τρόπο που συζητούμε άλλου είδους θέματα. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Για το θέμα αυτό λοιπόν υπάρχει κάτι που με ανησυχεί και έχει να κάνει με τον έλεγχο. Εγώ πιστεύω, πιστεύουμε τα μάλλα, την βιομηχανία, τον τομέα μπορούμε να ε, προσδώσουμε όλη την απαραίτητη εμπιστοσύνη έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν δοκιμές και να θέσουν στην αγορά το αποτέλεσμα των ερευνών τους γιατί αυτό αυξάνει την ποιότητα ζωής μας. Όμως ο έλεγχος ε, στον τομέα του ελέγχου είναι απαραίτητη θεμελιώδης η παρουσία του δημοσίου τομέα. Όταν μιλάμε για την υγεία έχουμε και ένα ισχυρό μέσο ελέγχου γιατί έχουμε το δίκτυο των νοσοκομείων και των γιατρών που μπορούν συνεχώς να χορηγούν στοιχεία με αρκετά χαμηλό κόστος. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλάμε επί της ουσίας για τον έλεγχο και ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε με συμμετοχή του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν, η κυρία Λίντστρομ, έχει το λόγο. ο κύριος. Α, Στέφαν Φιούρι. Α, α, έχω τον λάθος κατάλογο μπροστά μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω τώρα. Ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό της έκθεσης και για τη συνεργασία. Θα ήθελα να φερθώ σε πέντε σημεία, σας σύντομα, εν ώψη και των ε, παρεμβάσεων που ακούστηκαν. Καταρχήν η έγκριση. Η Κομισιόν δεν σκοπεύει με την πρόταση αυτή, μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα, οι όροι έγκρισης να μειωθούν λόγω του ότι θα υπάρχει μία άδεια εμπορία υπό όρους. κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σαφής οι κανόνες εδώ και οπωσδήποτε δεν σκοπεύει το... η Κομισιόν να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που θέλει να πετύχει η Κομισιόν με αυτή την πρότασή της είναι οι αρχές έγκρισης ζητούν περισσότερες πληροφορίες και να μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αρχή έγκριση στην εθνική διαδικασία να δώσει μια έγκριση και μετά να ζητήσει και άλλες πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι μπορεί για επιστημονικούς λόγους να χρειαστούν συμπραγματικές πληροφορίες. Λοιπόν, το τονίζω ότι δεν προτίθεμε θα να μειώσουμε τις απαιτήσει για την έγκριση ενός φαρμακευτικού διασκευάσματος. Δεύτερον, η κοινοποίηση στην τράπεζα δεδομένων. Θεωρούμε ότι σε μια ιστορική αγορά σήμερα δεν έχει κανένα νόημα για το ίδιο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, να γίνεται κοινοποίηση σε διάφορες εθνικές ε, τράπεζες δεδομένων και μάλιστα μια που έχουμε μια ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων που λειτουργεί, ίσως πρέπει να βελτιωθεί. Και μάλιστα όταν αυτό αφορά κάποιο φάρμακο που διατίθεται σε όλη την Ένωση ενδεχομένω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος μέλος ε, αποκλείεται από τι πληροφορίε, αλλά ότι μπορεί να πάρει πληροφορίε από την κεντρική τράπεζα δεδομένων. Τρίτο σημείο. Ε, η ενημέρωση μέσα στη συσκευασία που αναφέρθηκε για την ε, ε, ενημέρωση των ασθενών. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα και η, ο κίνδυνος. Αυτό το φυλάδιο λοιπόν είναι πολύ πιο σημαντικό από την οδηγία χρήση κάποιου παιχνιδιού. Γιατί εδώ θα πρέπει να αναφέρεται και ο κίνδυνος. Και η αποτελεσματικότητα. Και τα δύο. Η πρότασή μας προσπαθεί να λάβει υπόψη και τις δύο πτυχές. Να συνενωθούν σε μία ευρεία δήλωση και πιστεύουμε ότι είναι επικίνδυνο να φέρομαστε μόνο στον κίνδυνο στα φυλάδια αυτά ενημέρωση. Γιατί τότε το αποτέλεσμα είναι ότι ίσως ξεχνάμε το θέμα της αποτελεσματικότητας. Το κάτω-κάτω υπάρχει κάποιος λόγος γιατί ο γιατρός δίνει μια συνταγή για κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο. Δεν είναι μονάχα για να τρομάξει ο αλλά γιατί τους βοηθήσει. Τρίτο, διαφάνεια. Θα πρέπει να μπορεί η κοινή γνώμη να έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες. Θα πρέπει όμως να δούμε κατά πόσον είναι λογικό να ζητάμε όλες τις πληροφορίες σε αυτή την τράπεζα δεδομένων που να είναι ανοιχτή για όλο το ευρύ κοινό, γιατί αυτό ίσως είναι αντιπαραγωγικό. Και αυτό επιλέξαμε εμείς κάποια διατύπωση που επιτρέπει ευελιξία. Τέλος, τελευταίο σημείο που αφορά τη χρηματοδότηση. Πράγματι, η πρόταση για τον κανονισμό δίνει τη δυνατότητα κάποιες δραστηριότητε φαρμακοπαγρύπνηση να συσχετίζονται με έναν τέλος που θα καταβάλλεται από την φαρμακοβιομηχανία. Δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν επιδράσεις στις δραστηριότητες της ε, υπηρεσίας ε, προς την κατεύθυνση της βιομηχανίας μου φαίνεται λογικό, δεν θα πάω το αυτοκίνητό μου για το τεχνικό έλεγχο, πληρώνω ένα τέλος. Κανένας δεν λέει ότι επειδή έχω πληρώσει κάτι δεν γίνεται ο ελέγχος όπως πρέπει. Όχι. Ε, από εκεί που προέρχομαι εγώ πρέπει να πληρώσω ένα τέλος για να πάω στο δικαστήριο. Αλλά εγώ δεν άκουσα ποτέ κάποιο να λέει ότι αυτό το τέλος έχει επίδραση στην απόφαση του δικαστηρίου ή άμα πάω στην κρατική βιβλιοθήκη πρέπει να πληρώσω ένα τέλος, παρόλα αυτά το βιβλίο που δανείστηκα πρέπει να το πω πίσω, δεν μπορώ να το κατακρατήσω. Εκτός αυτού τέτοια τέλη υπάρχουν και σε άλλους τομείς και θα μπορούμε να θεωρήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται που δονεί η υπηρεσία να εξαρτηθεί γι' αυτό από την βιομηχανία. Και αυτή η πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί οι τράπεζες δεδομένων είναι πάντα πιο ακριβές από ό,τι φανταζόμαστε στην αρχή. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για τη λειτουργία αυτή τη τράπεζα δεδομένων να υπάρχουν κάποιοι πόροι συγκεκριμένοι και όχι μόνο το... ο κοινωνικό προπολογισμό, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι, η φαρμακοβιομηχανία, στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια κύριε Ριβάζη θέλει να επανέλθει. Μάλιστα, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνου που σα παρέμβησαν και να ευχαριστήσω και την Κομισιόν τη δική σα παρέμβαση. Δεν θέλω να επιστρέψω ξανά στι λεπτομέρειε, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Αναφέρεται που συχνά το θέμα της ανεξαρτησία και το θέμα της ε, σύγκρουση συμφερόντων. Είδατε που έγινε μια τέτοια έρευνα στο Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με μια σύγκρουση ενδιαφερόντων για τον ΠΟΕ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ξεκάθαροι ποιος κάνει τι, ποιος πληρώνει γιατί, ποιος πληρώνεται γιατί τι πράγμα. Άμα περάσουμε σε αυτή την Επιτροπή Αξιολόγηση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εκείνοι που θα αξιολογούν ε, τις παρενέργειες δεν είναι άτομα που πληρώνεται από τη φαρμακοβιομηχανία. Και ξέρετε η απάντηση του είναι ότι δεν θέλησαν να δώσουν τα ονόματα εκείνων που όρισαν Μα δεν, δεν επιτρέπεται. Ήθελαν, λέει, να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των εμπειρογνωμόνων. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει τα άτομα που γνωμοδοτούν πάνω στις παρενέργειες να είναι εξάρτητοι και να δίνουν το όνομά τους. Το βιογραφικό σημείωμα επίσης, γιατί όχι. Τώρα, εγώ μπορώ να συμφωνήσω να υπάρχει ένα τέλος που να επιτρέπει να χρηματοδοτηθούν τα περιφερειακά και εθνικά ε, κέντρα και η τράπεζα δεδομένων. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν ένα ε, εργαστήριο πληρώνεται κατά 100% από κάποιο τέλος, είτε σας αρέσει, σας αρέσει, θα υπάρχουν κάποιοι που θα επισέλθουν εκεί και θα αναμειχθούν. Εγώ είμαι υπέρ της διπλής χρηματοδότησης. Γιατί, γιατί θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εμπλακούν στο γεγονός ότι υπάρχουν κέντρα φαρμακοεπαγρύπνησης στις χώρες τους. Και η Ευρώπη επίσης να εμπλακεί εκεί για να χρηματοδοτήσει από ευρωπαϊκή σκοπιά την φαρμακοεπαγρύπνηση. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι μια υπηρεσία όπως κάποια άλλη. Τώρα, για τα φυλάδια ενημέρωση. υπάρχει κάτι που προτείνεται για τα νέα ε, φάρμακα και γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι οι ασθενείς που είμαστε όλοι, όλοι κάποια στιγμή είμαστε ασθενείς και θα χρειαστούμε να πάρουμε κάποια φάρμακα. Θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Ότι αν παίρνουμε ένα καινούριο φάρμακο, αυτό το φάρμακο δεν ε, έχει ε, Γι' αυτό το φάρμακο δεν υπάρχει πολύ μακρά πείρα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν πολύ, πολλά στοιχεία από πολλά χρόνια. Κατόπιν. Αναφέρομαι στο άρθρο 21 για να είναι σαφέ ότι πρώτοι για την εξαίρεση εξαίρεση. Τα φαρμακευτικά εργαστήρια τείνουν να πιέζουν τι άδειε αυτέ για να περάσουν στην διάθεση στην αγορά. Εμείς βέβαια δεν έχουμε σαν στόχο να τους πλουτίσουμε. Καθόλου είμαστε για να προστατεύσουμε την υγεία των ασθενών. Θα έχουμε λοιπόν το, την καλή μέση οδό. Σα παρακαλώ ξανά να διαβάσετε το άρθρο 21 για να δείτε ότι είναι αυτό που καλύπτει τι ε, ανησυχίε μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. 3 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Αυτό για πληροφορήσή σα. Περνάμε στο σημείο 17, ψευδεπίγραφα φάρμακα. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Σαρτόρη. Έχετε το λόγο κύριε Σαρτόρη. Πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τελικά μετά από πολλές ε, αναβολέ, ε, έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την οδηγία, για την πρόληψη ε, της κυκλοφορίας ψευδιοπίγραφων φαρμάκων στην ομιμελισίδα η παρουσία ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη φάρμα θρησκευτική ελισίδα αποτελεί πραγματική απειλή σε όλο το ευρωπαϊκό σύστημα γιατί υποσκάπτει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ποιότητα των φαρμάκων ε, που βρίσκονται στα φαρμακεία και σε οποιαδήποτε άλλα νόμιμα σημεία διανομή σήμερα. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι πολλούνται κάθε χρόνο ε, στην νόμιμη από την νόμιμη ελισίδα 1,5 εκατομμύριο κουτιά ψευδίγραφων φαρμάκων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν δεν αναλάβουμε αποφασιστική δράση, το νούμερο αυτό θα αυξηθεί το 2020 σε 40 εκατομμύρια ε, ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εντοπίζει με σαφήνεια τις αιτίες του προβλήματος, ε, όμως είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η ελισίδα διανομής, ε, οι υποχρεώσεις δεν είναι πάντοτε σαφείς, ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες κέρδους του τομέα που προσελκύει αυτές τις δυνατότητες παραχα και δίλια των φαρμάκων αν θέλετε και οι ποινές είναι αναποτελεσματικές ε, οι ή ελάχιστες. Ε, η πρόταση της Κομισιόν έχει κάποιες αδυναμίες που προσπαθήσαμε, επί των οποίων προσπαθήσαμε να παρέμβουμε με τροπολογίες που έχω παρουσιάσει 41, 41 τροπολογίες συνολικά. Εγώ προσπάθησα να ε, αναφερθώ στα θέματα αυτό. καταρθήν πρέπει να έχουμε ένα σαφή ορισμό για το τι εννοούμε με τον όρο ψευδεπίγραφο φάρμακο, τροπολογία 8 ένα ορισμό των ε, διάφορων ε, ε, υποκειμένων που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, έμποροι, παράλληλοι έμποροι και ενδιάμεση τροπολογία νέα. Ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω και το θέμα της ευθύνης των διάφορων εχομένων που συμμετέχουν στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Ο καθένας θα πρέπει να έχει μια άδεια για την επιτέλεση της εργασίας του και θα πρέπει να υπάρχουν βέλτιστε πρακτικές σε κοινοτικό επίπεδο. Θεώρησα λοιπόν απαραίτητο να ενισχύσω το θέμα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων γιατί αυτό είναι το μόνο πραγματικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας Αφενός ε, σκέφτηκα να προτείνω την ε, διαγραφή ε, της πιστοποιημένης οντότητας γιατί θεωρώ ότι αποδυναμώνει το σύστημα και δεν είναι κάτι χρήσιμο. Σύμφωνα με πρόταση της Κομισιόν θα μπορούσε να κάνει τις επιθεωρήσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να εγγυηθεί την ποιότητα του προϊόντος. Αυτή ε, αυτό το εγχείρημα σήμερα γίνεται χωρίς ε, ιδιαίτερο πρόβλημα από την ίδια την επιχείρηση παραγωγό ε, όταν, αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβλέψουμε μια νέα οντότητα θα ε, δυσκολίε δυσκολίες χωρίς κανένα πλεονέκτημα αφετέρου. Θεωρώ θεμελιώδες έτσι όπως ζητήθηκε και από γραπτή δήλωση που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών να καταστήσουμε γενικές το επιθεωρήσεις των ε, εξωτερικών εγκαταστάσεων παραγωγής προκειμένου να έχουμε εγγύσει για την ποιότητα και των δραστικών ουσιών και των φαρμάκων τα οποία είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε την ίχνηλασιμότητα. Ως προς ε, αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη εξηγήσει ε, παρά του, το έχει, παρά για το τι έχει γίνει ερώτηση πώς η Αμερικανική ε, ο Αμερικανικός Οργανισμός ε, μίλησε για έναν αριθμό 714 τέτοιων εξωτερικών εγκαταστάσεων, ενώ το έγγραφο που συνοδεύει αυτήν την οδηγία μιλά για 15 έως 20 χιλιάδες, ε, λέγοντας επομένως ότι είναι αδύνατο να γενικεύσουμε τους ελέγχους. Προκύπτει λοιπόν ότι μία συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός μικροκύκλου χωρών, όπως είπα η Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδά, με χώρες με τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, θα ε, μας διευκόλυνε να έχουμε τριετή τι έλεγχο σε κάθε εγκατάσταση, εξωτερική εγκατάσταση παραγωγής ε, φαρμάκων. Αν ε, βέβαια έχουμε έναν αριθμό από 5 έως 800 για να γίνει ε, αυτό το έργο θα αρκούσαν 40 επιθεωρητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να κλείσω, αναφέρθηκα και σε μία σειρά άλλων θεμάτων το εμπόριο μέσω του διαδικτύου. Έχουμε τροπολογίες 1.28.41 ε, και τα φάρμακα που πολλούνται απευθεία από τον παραγωγό στο νοσοκομείο που χορηγεί στον ασθενή το φάρμακο, τι κυρώσει το παράλληλο εμπόριο ή ε, προθεσμία της θέσης ισχύω της οδηγίας. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε το χρονικό διάστημα. Ε, έχουμε ως καταλεκτική ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, για την κατάθεση τραπολογιών. Εδώ λοιπόν εγώ ήθελα να διευκρινίσω κάποια δευτερεύοντα θέματα. Να προσθέσω όμως ακόμη και κάτι που αφορά τα έκδοχα. Πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα να εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέλτιστες πρακτικές παρασκευής έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ποιότητα και αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων και να λαμβάνουμε υπόψη ε, την ίδια τη φύση του εκδόχου και να λάβουμε υπόψη την περίπτωση όπου δεν έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα οι ουσίες αυτές. Επίσης, ε, να αναφερθώ ότι στις 13 ε, Νοεμβρίου ε, παρουσίασα, κατέθεσα μία γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μάθω πώς τα δεδομένα της Κομισιόν μιλούν για έναν αριθμό εγκαταστάσεων που παράγουν δραστικές ουσίες στο εξωτερικό από 15-20.000 ενώ ο Αμερικανικός Οργανισμός μας λέει ότι είναι 714. Η απάντηση ήταν ότι στη μελέτη αντικτύπου που οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται προέρχονται από τη ΣΕΦΙΚ, από τη Χημική Βιομηχανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το ότι αυτά τα δεδομένα αμφισβητούνται από τη Χημική Βιομηχανία. Εγώ έκανα αυτή την επαλήθευση και πρέπει να πω ότι και Ευρωπαϊκός, συγγνώμη, και η ίδια η ΣΕΦΙΚ αλλά και ο Αμερικανικός Οργανισμός συμφωνούν στο ότι ο αριθμός αυτών των εγκαταστάσεων δεν ξεπερνά σήμερα τις 800 και επομένως ε, μπορεί να εφαρμοστεί ε, αυτό που θέλουμε εμείς, δηλαδή η έλεγχη και επιθεωρήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντα έχει το λόγο. Um, thank you, um, and... Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και για τα σχόλιά της, αλλά και για τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο εκπώνησα την έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της ε, βιομηχανίας και των μεγάλων φαρμακευτικών ε, εταιριών μέχρι και τους ε, φαρμακοποιούς για το επίπεδο πληροφοριών που μας έδωσαν για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η βιομηχανία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όντως, πολλοί που εργάζονται στα ιατρικά επαγγέλματα έδωσαν εσωτερικές πληροφορίες για το πόσο, πόσο σημαντικό το θεωρούν αυτό. Εγώ είμαι παντρεμένη με γιατρό που ε, δίνει συντα, συνταγογραφή ε, φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έχω κάποια ίσως σημασία σχόλια που θέλω να κάνω και ίσως να υποβάλω και κάποιες τροπολογίες. Το πρώτο, τροπολογία 28. Πολύ σημαντικό θέμα για την ε, ευαισθητοποίηση του κοινού. Η δική μας εμπειρία από το Ρωμανό Βασίλειο λέει ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει έχει, έχει κάποιες, εκπονήσει κάποιες πολύ επιτυχημένες διαφημιστικές εξτρατείες για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Τώρα, ό,τι αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση, υπάρχει μεγάλη πίεση εκεί και όταν ο, ιδιωτικός, τομέα θέλει να χρηματοδοτήσει αυτές τις εξτρατείες, ίσως καλό θα ήταν να υπάρχει μια διατύπωση να γίνονται δηλαδή οι ε, ε, εξαρτίες αυτές, ε, να, να χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα και να υπάρχει ίσως υποπτή από το κράτος μέλος, από τις κρατικές αρχές. Ίσως κάτι τέτοιο να βοηθούσε να περάσει το μήνυμά μας. Δεύτερον, έλεγχη, εποπτεία. Συμφωνώ. Η εποπτεία είναι πολύ σημαντική και ευχαριστώ την εισηγητρία για την δουλειά που έκανε ό,τι αφορά το πόσοι ε, έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται. Γνωρίζω βέβαια ότι δεν θα πρέπει κατά ανάγκη να περιμένουμε από τις τρίτες χώρες να υποχρεούνται να έχουν υψηλότερο ε, επίπεδο ε, καθεστώ, υψηλότερο επίπεδο ελέγχων από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ζητήσουμε κάτι τέτοιο, αυτό θα, μπορέ, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προστατευτισμός και να έχει σημαντικά ε, συνέπειες. Οπότε ας το δούμε πολύ προσεκτικά το θέμα των καθεστώτων ε, των ελεκτικών και ας μην ε, επιβάλλουμε αχρία στους ελέγχους στις τρίτες χώρες, ώστε ο κίνδυνος και τα ωφέλη που θα λάβουμε να είναι σε ίσο επίπεδο. Τώρα, για το, επίπεδο, για το πεδίο εφαρμογή και το αν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μόνο συνταγογραφημένα φάρμακα ή μη συνταγογραφημένα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν φάρμακα που δεν χρειάζονται συνταγογράφηση. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις κάτω χώρες, υπάρχει αρκετά φιλελεύθερο σύστημα που μπορεί κανείς να πάει και να αγοράσει ένα πακέτο ασπιρίνες, ας πούμε ή παναντόλ από το γωνιακό του φαρμακείο. Αν τώρα πάμε στα πολύ βασικά φάρμακα που δίδονται χωρίς συνταγοράφηση και, και τα υποβάλλουμε στις ίδιες απαιτήσει ασφάλειας για αυτά που έχουμε που είναι πιο ακριβά και που χρειάζονται συνταγογράφηση, τότε μπορεί να υπάρχουν μεγάλες συνέπειες μεταξύ των κρατών μελών, γιατί οι καταναλωτές μπορούν σε κάποια κρατημέλη να αγοράσουν αυτά τα βασικά φάρμακα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε ας έχουμε μία προσέγγιση πάλι με βάση τον κίνδυνο. Αν δηλαδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για κάποιο φάρμακο να είναι ε, ψευδεπίγραφο, ας έχουμε έναν κατάλογο τέτοιων φαρμάκων. Ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος για να προχωρήσουμε. Κατά τα λοιπά, ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε και θα σας υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες και ευχαριστώ που έχετε λάβει υπόψη και αυτές που έχουμε ήδη υποβάλει. Ο Να συγχαρώ την ε, συνάδελφο για τον τρόπο με τον οποίο διχειρίστηκε το θέμα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ καλέ οι τροπολογίε. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την πρώτη, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι το, πρώτο, το βασικό πρόβλημα. Ε, κάτι που έλειπε δηλαδή μέχρι στιγμή. Ίντερνετ. Το ίντερνετ και το εμπόριο από το ίντερνετ είναι ένα βασικό, μια βασική πηγή τέτοιων ψευδοεπίγραφων φαρμάκων. Το ΙΤΡΕΝ μέχρι στιγμή δεν, έχει, δεν αναφερόταν στον, στην πρόταση και νομίζω ότι χρειάζεται ένα διπλό διπλός ε, συνδυασμός, όπως είπε και η κυρία Φόρτ. Μιλούμε για την ευαισθητοποίηση των ασθενών, ώστε να γνωρίζουν ότι όταν παίρνουν από το, ε, από το ίντερνετ ένα ε, μη στεγογραφημένο ε, φάρμακο ε, έχουν, υπάρχει ο κίνδυνος να, μην, να είναι ψευδεπίγραφο, οπότε χαίρομαι που η εισηγήτρια, και βλέπω ότι και οι υπόλοιπε ε, ομάδες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Συμπεριλαμβάνει το ίντερνετ και το υποστηρίζω στεναρά. Η Κομισιόν μέχρι στιγμή είχε κάποιε αμφιβολίε ω προ αυτό. Το γνωρίζω γιατί δεν, ε, είναι, δεν επιτρέπεται σε κάθε χώρα το εμπόριο μέσω ίντερνετ. Αλλά αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό, θέμα ιστορική αγορά. Πέρα από αυτό, το θέμα των ε, χαρακτηριστικών ασφαλεία που αναφέρονται εδώ. Θα πρέπει να αποφύγουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, το υψηλό κόστο, ποιο θα το αναλάβει, το υψηλότερο κόστος. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα, νομίζω εγώ, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις, ε, τις αποδόσεις που έχουμε και να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχει ανιχνευσιμότητα. Ε, χρειαζόμαστε δηλαδή σαφήνεια από πού προέρχεται αυτό το προϊόν. Αλλά αυτό που δεν θέλουμε είναι ο ασθενής, ο πελάτης, στο τέλος της αλυσίδα να συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα. Α, θα πρέπει το σύστημα να τελειώνει στο φαρμακείο, γιατί αλλιώ υπάρχει θέμα ε, προστασία δεδομένων. Η ανιχνευσιμότητα θα πρέπει να σταματάει σε ένα σημείο και θα πρέπει να γίνεται αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση ε, να μην έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ε, των ε, ασθενών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας που στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει εκπονήσει μια εξαιρετική έκθεση. Όντως και οι οργανώσεις καταναλωτών και η βιομηχανία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Θα ξεκινήσω με κάποια σημεία που τα υποστηρίζω πλήρως. Και τα ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Το ίντερνετ είναι ένα σημαντικό τμήμα της έκθεσης ε, και εκεί είναι η πύλη για το σύστημα ε, προμήθειας της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει νομίζω συμφωνία ως προς αυτό ότι θα συμπεριληφθεί πια στην οδηγία το ίντερνετ. Επίση, πολύ καλό είναι το γεγονός ότι η κυρία ε, Σαρτόρη κάνει διαχωρισμό μεταξύ εμπορευόμενων ε, και ε, χρηματο... μεσητών. Συμφωνώ ότι όντως θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αρχές σύμφωνα με τις οποίες να κινούμεθα και είτε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, είτε θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές καθεστώς, να υπάρχουν δηλαδή σαφείς ε, πρακτικές. Έρχομαι τώρα στο σημείο με το οποίο δεν νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Είναι σημαντικό να δούμε το κόστος του προϊόντος για τον καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτής είναι αυτός που θα καταβάλει το κόστος γιατί υπάρχουν ε, και θέματα έξτρα ελέγχων κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πολύ καλό σύστημα ελεγκτικό ήδη και αυτό το σύστημα που εμείς εφαρμόσαμε πρόσφατα λειτουργεί. Αλλά μπορεί να μην λειτουργεί σε όλες τις χώρες. Αλλά δεν θα... Δεν σημαίνει ότι αν αλλάξουμε τα πράγματα φορτώνουμε πάρα πολύ το σύστημα. Μήπως θα πρέπει απλώς να το τροποποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί για όλους. Γιατί δεν συμφωνώ καθόλου ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύστημα ε, ελέγχων, ακόμη πιο λεπτομερές ε, από αυτό που έχουμε. Η υγεία των ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να γίνονται Έλεγχη κάθε τρία χρόνια όλων των κατασκευαστικών ε, των φαρμακοβιομηχανιών, ε, είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Ακόμη και αν γίνει πολύ σκληρή δουλειά, μόλις 8% ε, των ελέγχων ετησίως θα μπορεί να γίνει. Οπότε δεν γίνεται να ελεγχθούν όλα τα εργοστάσια. Θα χρειαστούν 13 χρόνια. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ας βρούμε έναν εφικτό τρόπο για να προχωρήσουμε. Όπως και η συνάδελφος, ας ε, διατηρήσουμε, ας έχουμε υπόψη μας το ε, πεδίο εφαρμογή αυτής της πρότασης, να αποφύγουμε τα ψευδεπίγραφα, όχι να επιβάλλουμε άπειρους ελέγχου. Οπότε, ας μην χρησιμοποιούμε κανόνι για να σκοτώσουμε κουνούπι, Ας δούμε τι είναι εφικτό στα πλαίσια αυτών των ε, συστημάτων ελέγχων που έχουμε και ας προχωρήσουμε έτσι. Επίσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των συνταγογραφημένων και των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων. Η κυρία Ματίας το είπε στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση μετά από τα πέντε χρόνια για να δούμε αν τα μη συνταγογραφημένα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Στην ε, περίπτωση ε, τώρα δεν, ε, δεν συμπεριλαμβάνονται και το υποστηρίζω αυτό. Επίσης, μιλούμε για το πεδίο εφαρμογή και μιλούμε για τις κυρώσεις και υπάρχει ένας κάποιος, ένα κάποιο πρόβλημα με τους ορισμούς. Τι είναι το ψευδεπίγραφο προϊόν. Και σας παραθέτω από αυτά που λέει η ΠΟΗ, ένα ε, προϊόν το οποίο ενσυνείδητα έχει, είναι ψευδεπίγραφο, είναι, έχει, είναι κύβδηλο. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, σύντομα, ο κύριος Φούριν και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία-τέσσερα πραγματάκια να πω κι εγώ. Για τον ορισμό του ψευδεπίγραφου φαρμάκου. Είναι σημαντικό να είναι σαφής ο ορισμός, να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε εμείς όταν λέμε ψευδεπίγραφο. Δεν μιλούμε για πνευματική ιδιοκτησία εδώ, για αγορές και τέτοια. Μιλούμε για, ασχολούμαστε με τελείως διαφορετικό θέμα ούτε για διπλώματα ευρεσιτεχνία μιλάμε. Οπότε ο ορισμό για τον οποίο συζητούμε εδώ πάει προ σωστή κατεύθυνση. Δεν μιλούμε για παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνία. Μιλούμε για ένα προϊόν το οποίο δεν ε, έχει έγκριση, δεν είναι εγκεκριμένο. Αυτά για τους ε, ορισμούς καταρχήν. Για τους ελέγχους τώρα. Όντως, το σύστημα τώρα βασίζεται στο ότι ο παρασκευαστής είναι, έχει έναν εγκεκριμένο ε, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που ε, ελέγχει την ποιότητα των φαρμάκων. Αυτή είναι η βάση του συστήματος και προς το παρόν οι έλεγχοι δεν καλύπτουν τα πάντα, δεν καλύπτουν όλους τους προμηθευτές, ούτε αυτό αναφέρεται και στην οδηγία. Καμιά φορά ακούγεται ότι αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται παντού, για όλους τους προμηθευτές, σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε της άποψης ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Προς το παρόν τουλάχιστον με τους πόρους που έχουμε. Οπότε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα όσο έχει, αλλά παρόλα αυτά να ενισχύσουμε τους ελέγχους. Αυτό ναι αλλά να αποφύγουμε καταστάσεις όπου ένας παραγωγός ε, μπορεί να εισαγάγει ενεργές ουσίες στην ε, Ένωση ε, μόνο αφού ελεγχθεί. Οι ενεργές ουσίες μόνο σε τρίτες χώρες παράγονται προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αριθμητικά στοιχεία, εκεί υπάρχουν τελείω διαφορετικές απόψει. Αν δούμε τους καινούργιους αριθμού, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Καταρχήν, τυπικά δεν ε, ελέγχονται ε, εγκαταστάσεις αλλά γραμμές παραγωγής. Κάποια πολύ, μερικές, ε, μερικές εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες αποτελούνται από πολλές γραμμές παραγωγής. Ελέγχουμε λοιπόν τις γραμμές παραγωγής. Και δεύτερον, τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει ενεργή ουσία σε κάποιες χώρες, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξει ε, μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τον ορισμό και αν επιβάλλουμε εμείς έναν ορισμό μπορεί να καταλήξουμε να ελέγχουμε πολύ λίγους τελικά παρασκευαστές. Οι ελεγκτές που δουλεύουν για μας και που βρίσκονται εδώ στην Ευρώπη ελέγχουν περίπου 400-500 εγκαταστάσεις. Και είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλοί περισσότεροι παρασκευαστές και στη δική μας αξιολόγηση επιπτώσεων θεωρούμε ότι μπορεί να φτάσει τους, τις 20.000 ε, γραμμές παραγωγής ο αριθμός αυτός, σε τρίτες χώρες τουλάχιστον. Οπότε θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να επιβάλλουμε υποχρεωτικούς ελέγχους στους πάντες. Σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, πρώτο τελευταίο σημείο, είμαστε ανοιχτοί για νέες δυνατότητες, για εξτρατείε ε, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι διατάξεις ε, που αφορούν το εμπόριο ε, στο ίντερνετ είναι τελείως διαφορετικές στα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη ε, το απαγορεύουν πλήρω, κάποιοι, κάποια κρατημέλη το επιτρέπουν εν μέρη. Ε, υπάρχουν διάφορες... Ε, είναι κλιμακωτά τα πράγματα σε αυτό. Και εφαρμογή και σχετικές διατάξεις. Και εδώ το ίδιο ισχύει όπως και με του ελέγχου. Έτοιμά μα α είμαστε ρεαλιστές. Μέσα σε λίγους μήνες δεν γίνεται να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα ελέγχων. Μέσα σε λίγους μήνες μπορούμε να προβλέψουμε κάποια φάρμακα που να, και να τα ελέγξουμε με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε έτσι πιο μακροπρόθεσμα. αλλά θα συμφωνήσουμε ότι όντως αυτό πρέπει να γίνει ως το δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτόρη θέλει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους. Συνεισφέρουν τα μάλα στο έργο που θα παρουσιάσω στη συνέχεια και πραγματικά με εξυπηρετεί στην παρουσίαση των Υπουργείων. Ευχαριστώ. 3 Φεβρουαρίου προθεσμία για υποβολή ε, τροπολογιών. Το είπε και η κυρία Σαρτόρη. Πάμε στο σημείο 18. Κινητοποίηση των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση τη μετάβαση προ μια ενεργειακά αποδοτική ή οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε νομοδότηση που εκπανώ και για την οποία σήμερα θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετίζεται με δύο νομοθετήματα της Κομισιόν, μια ανακοίνωση του περασμένου έτους ε, και μία σύσταση της Επιτροπής ε, πάλι του περασμένου έτους ε, όπου αναφέρονται κάποιες προτάσεις και προσαρμογές. Μιλάμε για τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, ICT, για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Δύο λόγια, πολύ σύντομα, για να πλαισιώσω τη γνωμοδότησή μου, τη γνωμοδότησή μας που θα παρουσιάσουμε εμείς ως Επιτροπή στην πιο γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτεύξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων η Ευρώπη για να διατηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για το 2020 και ενεργειακού χαρακτήρα κυρίως θέλει με, αυτή την, με αυτό το νομοθέτημα αλλά και με άλλα που έχουν ήδη υιοθετηθεί να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερες δεσμεύσεις ε, για την ενεργειακή εξοικονόμηση και κυρίως εδώ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι λοιπόν εδώ εισάγονται κάποιες καινοτόμες παρεμβάσεις σε σχέση ε, με άλλα που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή μας γιατί θέλουμε συγκεκριμένα επί της ουσίας να τονίσουμε τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και να δούμε πώς, και αυτά είναι τα δύο κυρία στοιχεία, πώς ο τομέας αυτός ε, μπορεί στη δική του δραστηριότητα, δηλαδή στη βιομηχανική παραγωγή του τομέα τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών, να ε, μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ε, για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο τομέας αυτός τεχνολογιών στο εσωτερικό του και κατά πόσο οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω και να εισαχθούν στο βιομηχανικό τομέα και να αποτελέσουν ένα στοιχείο για την επίτευξη πιο υψηλών στόχων ενεργειακή αποθετικότητα. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μια καταλητική λειτουργία, δηλαδή τα προϊόντα αυτά θα είναι προϊόντα καταλύτες ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και επίσης έχουμε και ε, ένα καινοτόμο χαρακτήρα γιατί πολλές φορές ε, θέτουμε στόχους αλλά τελικά δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτές και αν έχουμε αυτά τα μέσα μέτρησης αυτά τα συστήματα, τις συσκευές μέτρησης, ε, τότε ε, μπορούμε να ε, έχουμε μία σειρά δεδομένων. Όμως θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να είναι συγκρίσιμα, γιατί διαφορετικά χάνουμε την αξιοπιστία μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέρα από αυτό έχουμε και απώλεια αποτελεσματικότητας, γιατί δεν πετυχαίνουμε το στόχο. Πρόκειται λοιπόν εδώ για ένα νομοθετήμα που θέλει να τονίσει την ενεργειακή απόδοση. Και όπως ε, σας είπα στις διατάξεις ε, αυτές ε, και στη σύσταση θέλουμε να τονίσουμε τη δυνατότητα επαλήθευσης του πόση ενέργεια καταναλώνουμε και πόση εξοικονομούμε και ε, υπάρχουν ε, και όργανα μέτρηση σε πραγματικό χρόνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές έτσι ώστε να διορθώσουν λαθασμένες ε, συμπεριφορές ενδεχομένως. Μπορούν λοιπόν να συνεισφέρουν εδώ αυτά σε δύο τομείς, τεχνολογίες, σε ό,τι αφορά καταρχήν τις υποδομές, τις κατασκευές αλλά και τις μεταφορές και πολλές φορές όταν ε, αναφερθήκαμε στην ενεργειακή αποδοσία των κτηρίων, αναφερθήκαμε στα θέματα αυτά. Εδώ θέλουμε να πάμε όμως ε, λίγο παραπέρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας ε, στα κτίρια και στις κατοικίες φτάνει το 40% της κατανάλωσης, 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές φτάνουν στο 25% περίπου. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι τομείς κατανάλωσης. Ε, έτσι λοιπόν ε, εδώ ε, στον τομέα των κατασκευών και στον τομέα της διαχείρισης των κατασκευών θέλουμε και στον τομέα των μεταφορών θέλουμε να δώσουμε έμφαση για να δούμε πώς τους τομείς αυτούς οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να συνεισφέρουν για να περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση. Και τελικά θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο της ενεργειακής κατανάλωσης. Και κάτι ακόμη που είναι ενδιαφέρον κατά την άποψή μου και το υπογραμμίζω αυτό στη γνωμοδότηση είναι ότι εδώ θα δράσουμε στη ζήτηση, επί της ζήτησης. Πώς μπορούμε λοιπόν να εισαγάγουμε μέσα και τρόπους έτσι ώστε και στο επίπεδο της ζήτησης θα έχουμε κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν και οι ίδιοι οι καταναλωτέ να μειώσουν την κατανάλωσή του και να περάσουν στην αποδοτικότητα. Δηλαδή δεν λέμε να καταναλώνουν λιγότερο και να ζουν χειρότερα, αλλά να ζουν με τον ίδιο τρόπο, απλώ χρησιμοποιώντα λιγότερη ενέργεια, γιατί θα υπάρχει ενεργειακή απόδοση. Ε, μιλάμε για τις οικογένειες, για τον μεμονωμένο καταναλωτή, για τους θεσμικούς καταναλωτές, δηλαδή τις δημόσιες οντότητε τους δημόσιου οργανισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις. Έχουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον κόσμο της παραγωγής. Και εδώ παρουσιάζονται κάποια πρώτα μέτρα στην νομοθεσία και εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο παραπέρα πιο εις βάθος γιατί μιλάμε για μονομένους καταναλωτές ε, και να το χάρη εδώ σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι έξυπνοι μετρητέ από τους καταναλωτές για να μπορέσει ο καταναλωτή να χρησιμοποιεί καλύτερα την ενέργεια αλλά έχουμε κατά νου και τους θεσμούς να το χάρη όταν έχουμε ε, δημόσιους ε, διαγωνισμούς, δημόσιες συμβάσεις να τίθεται όροι για το τι μπορούν να κάνουν και οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά ε, να μιλάμε και για τις υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και σε άλλους στρατηγικούς τομείς δημόσιων υπηρεσιών. Πάρα πολλά θα μπορούσαν να γίνουν ε, από την πλευρά των δημόσιων θεσμών χρησιμοποιώντας αυτές ε, τις νέες τεχνολογίες. Και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα υπάρχουν ε, καλές πρωτοβουλίες ε, για περισσότερη παραγωγή. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για ορισμένες χώρες της Ευρώπης και για τη δική μου που υπάρχουν ε, πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και φυσικά αυτό έχει επίπτωση και στο κόστος και στην κατανάλωση πρώτων υλών. Έτσι λοιπόν, από όλες αυτές τις προτάσεις τα έγγραφα τη Κομισιόν υπάρχουν πέρα από όλε αυτές τι προτάσει, υπάρχουν και ορισμένε δεσμεύσει και ορισμένε προθεσμίες. Στο πρώτο έγγραφο της Κομισιόν ε, υπάρχει ένας ε, πίνακας, αναφέρονται τα μέτρα, το χρονοδιάγραμμα και τα διάφορα στάδια. Ε, όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ γενικόλογα όλα αυτά και υπάρχει και απόκληση μεταξύ των διαφορών εγγράφων. Εγώ θα πρότεινα στην Κομισιόν να εργαστεί λίγο περισσότερο επί των πτυχών αυτών. Γιατί, εντάξει, καλό είναι να θέτουμε στόχους, αλλά πρέπει να πούμε και πώ θα τους πετύχουμε. Λόγου χάρη, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερα το εξή αν λέμε κάθε κράτο μέλος Ε, τελικά πρέπει να κάνει κάποια δήλωση προθέσεων. Ε, δηλαδή πρέπει να απευθυνθεί στις βιομηχανίες, ε, στον τομέα τεχνολογικών πληροφοριών και στον τομέα των μεταφορών. Και όλοι αυτοί πρέπει να αποφασίσουν από κοινού για τις προθέσεις τους, για τη βούλησή τους να υιοθετήσουν σχέδια και εναλλακτικά μέτρα. Νομίζω ότι αυτά είναι ορθά, ορθές ιδέες, αλλά πρέπει να διαρθρωθούν καλύτερα στο τομέα των ταυπιών Ζητείτε ζητείται κάθε χώρα μέσα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ε, να υπάρχει αυτό ο πίνακα και η κοινή δήλωση προθέσεων και να υπάρχει και ένας οδικό χάρτη, δηλαδή να πει κάθε χώρα ε, τι θέλει να μελετήσει για να, και να υιοθετήσει για να φτάσει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ξέρετε ότι και η στρατηγική της Λισαβόνα σε μεγάλο βαθμό απέτυχε γιατί δεν είχε καθοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος επίτευξης των στόχων. Και στη συνέχεια κάθε κράτος αναλαμβάνει τις συνέπειες για το τι κάνει και τι δεν κάνει. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καλύτερο τρόπος ε, να διαρθρώσουμε αυτές τις προθεσμίες και υπάρχουν δύο λεπτά πρόεδρε. Να προσθέσω ότι για το δικό μου σχέδιο έκθεσης προτείνω η Κομισιόν μέσα σε αυτό το έτος να καταρτήσει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον ε, για τις ε, προθεσμίες, για όλα αυτά τα περάσματα στα διάφορα μέτρα και στους διάφορους τομείς. Και υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις, κάποιες υποχρεώσεις και θα ήθελα κυρίω να τονίσω στι υποχρεώσει που θα πρέπει να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί συνήθω αυτή είναι η πρώτη που δεν σέβεται τι υποχρεώσει που έχουν τεθεί. Και εδώ βλέπω ότι μπορεί να γίνει για πολύ καλή δουλειά στο πώς χρησιμοποιούν οι πολίτες τις δημόσιες υπηρεσίες αυτή η τυποποίηση ε, των ε, μέτρων επίσης είναι σημαντική γιατί πολλές φορές δεν κατορθώνουμε να έχουμε ε, τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάποιο σε έντυπε συζητήσει είπε να θέσουμε το θέμα τη ενεργειακή αποδοτικότητα ω υποχρεωτικό στόχο στου διάφορου τρόπου εργασία μα. Φυσικά αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, είναι ιδιαίτερα γενική η πρόταση αυτή και θα πρέπει να συζητηθεί. Σταματώ εδώ, λέγοντας ότι ενδιαφέρομαι για όλες τις ε, συνεισφορές σας, γιατί θεωρώ ότι εδώ έχουμε κάποια ε, θετικά ε, νομοθετήματα και θα μπορούσαμε εμείς να συνεισφέρουμε για να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι και πιο αυστηροί. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, βέβαια. Στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές στρατηγικές που έχουν ονόματα πόλεων, εποχών του έτους. Στο μέτρο της ενέργειας έχουμε το 2020 που πρέπει να πετύχουμε σε 10 χρόνια. Αλλά το θέμα που συζητούν όλοι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα λέγαμε ότι είναι ένα θέμα πολύ σεξ. Ο πνευματική χρήση ενέργειας δεν είναι τόσο προκλητικό. Δεν συζητιέται τόσο πολύ γιατί δεν γίνεται τόσο κατανοητό. Πάρα αυτό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες οικονομίες αυτή η ανακοίνωση κομισιών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε οπωσδήποτε, γιατί η αποτελεσματική χρήση ενέργειας είναι το επίκεντρο που καταδεικνύει τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων του 2020 και πώς θα εκμεταλλευτούμε το ECT για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Αυτό τι σημαίνει. Αφενός γνωρίζουμε ότι μία οδηγία που θα έχουμε θέσει θα μπορέσει να μας βοηθήσει καλύτερα να ορίσουμε στόχους, να ορίσουμε ε, συντονιστές, να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας ή ηλεκτρικού, δηλαδή να αγοράζει κανένας ε, μια συσκευή που είναι σύμφωνη με ε, ένα καλύτερο πρότυπο χρήση ενέργειας ΑΒΓ, ξέρετε πώς είναι η ταξινόμηση αυτή. Το άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ε, εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι η χρήση του ICT e είναι τέτοια που να μπορεί να χρησιμοποιεί έξυπνες ε, μεθόδους καταμέτρησης. Οι εγκαταστάσεις smart δηλαδή όπως λέγονται που δίνει στον καταναλωτή την πληροφορία το πόση ενέργεια καταναλώνει κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Εγώ δεν έχω στο σπίτι μου και κανένα άλλο έχει νομίζω τέτοια εγκατάσταση. Έχω αυτή την μπαμπάλια μέθοδο που μετράει πόσα κιλοβάτ καταναλώνω ένα ευφυής μετρητής θα μπορεί όμως σε πραγματικό χρόνο να δίνει τις πληροφορίες στον καταναλωτή το τι ε, καταναλώνει κάθε στιγμή. Να μην χρησιμοποιεί σε κάθε μέρα τόσο πολύ ε, ενέργεια. Θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής να αγοράζει φτηνότερα το τον ηλεκτρισμό του, να πλένει ας πούμε, τα ρούχα του ή τα πιάτα του τη νύχτα και να εκμεταλλεύεται τις περιόδους αυτού της ε, χαμηλής ζήτησης. Αυτό που μας λείπει στην Ευρώπη είναι ότι δεν έχουμε κοινά πρότυπα, όπως είπε και η εισηγήτρια. Η εισηγήτρια προτείνει να εισαγάγουμε για τους ευείς αυτούς μετρητές αυτά τα κοινά ευρωπαϊκό πρότυπα. Μου φαίνεται ότι θα ήταν πολύ καλό, γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε την τεχνολογία αυτή πιο γλίγορα και να την εκμεταλλευτούμε πιο γλίγορα. Οι μετρητές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τέτοιου τύπου δίκτυα ενέργειας που να συμπεριλαμβάνουν και πιο καλές πηγές ενέργειας. Παραδείγματο χάρη, ε, η ηλιακή ενέργεια, όταν υπάρχει ήλιος, η αιωλική ενέργεια, αν φυσά ο Και ε, θα μπορέσουμε έτσι να γνωρίζουμε και τον, την πραγματική μας κατανάλωση. Όπως είπα, θα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να αναπτύξουμε αυτές τις ευφυείς τεχνολογίες. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν, ιδίως όσον αφορά αυτή την, αυτά τα ενιαία πρότυπα για τους μετρητές. Ευχαριστώ. Ποιος μας. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που μπορεί να ξέρει κανένας ότι εάν πάει μία φορά στο Google είναι σαν να αφήνει το φως αναμένο ώρες. Δηλαδή το ECT οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και θα πρέπει να φροντίσουμε τα τεράστια κέντρα ε, υπολογιστών που υπάρχουν λίγο πολύ παντού να ε, Θα μπορούσε να έχει κανένας πιο μικρές μονάδες, να τις δικτυώσει μεταξύ τους και έτσι να γίνει και μια πιο σημαντική οικονομία ε, ηλεκτρισμού. Δηλαδή η βιομηχανία θα πρέπει καταρχήν να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από την ίδια. Δεν πρέπει να συζητάνε για τους άλλους και να μην κοιτάνε τι κάνουν οι ίδιοι. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Μπορώ να συμφωνώ με συμφωνήσω με τον κύριο Καρίντς ότι οι κύριες εξοικονομήσεις από την ΕΣΕΤΕ θα γίνουν ε, όταν χρησιμοποιήσουμε ευφύης μετρητές. Σήμερα το κόστος παραγωγής είναι 70% ενέργεια, νερό και μόνο το 20-30% είναι το εργατικό κόστος για κάποια παραγωγή στην Ευρώπη. Και ένα από τα σημαντικότερα που θα μπορούμε να επιτύχουμε με το στόχους του 2020 θα είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και εκεί θα παίξει να και μπορούμε πολλά έτσι να πετύχουμε γλυγορά. Το άλλο είναι, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα ευφυή e e δίκτυα και τους ευφυείς e μετρητές, Smart Greek και Smart Meters. Υπάρχουν διάφορες με τι είναι ο ευφυής μετρητής. Αναφέρεται συχνά κανείς στην Ελ στην Ιταλία. Τι ήταν το πρόβλημα. Πολλοί δεν πλήρωναν τον ηλεκτρισμό στην Ιταλία και είναι προετοίμασε ένα ευφυή μετρητή χαμηλής τεχνολογίας που του μέρισε σε όλα τα νοικοκυριά για να βελτιωθεί ε, η αντιμετώπιση των Ιταλών όσον αφορά τους, την πληρωμή του λογαριασμού. Αυτοί οι ευφυείς μετρητές δεν μπορούν παρά να είναι ανοιχτοί ή κλειστοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πριν προσπαθήσουμε να βάλουμε ευφύς μετρητές σε κάθε νοικοκυριό θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε τι θα πρέπει να μπορεί να επιτύχει ένας ευφύς μετρητής. Να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή ένας τέτοιος μετρητής που εγκαθίσταται σήμερα να μπορεί σε 5-6 χρόνια να μετατραπεί για διαλειτουργικότητα. Κάτι άλλο. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν κίνητρα για τους καταναλωτές, για τους ευφυείς μετρητές. Γιατί? Γιατί καταρχήν η κατανάλωση στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγαλύτερη ε, από ότι στην Ευρώπη. Γιατί έχουν περισσότερη ηλεκτρική θέρμανση, κλιματισμό και ε, κακή μόνο στα σπίτια τους. Εκείνοι μπορούν να κάνουν πολύ, πολύ περισσότερες οικονομίες από ότι οι Ευρωπαίοι. Το κόστος που θα είχα, ούτως ώστε εκατομμύρια ηλεκτρικά πλυντήρια να ελέγχονται και να μπαίνουν σε λειτουργία μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Είναι πολύ πιο ακριβό το, το κόστος αυτό παρά εάν ε, τροποποιήσω 500 βιομηχανικές μονάδες ή 50.000 ΜΜΕ. Αυτά είναι πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο φθηνά να οργανωθεί από ότι 50-500 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη με τα πλυντήριά τους τα ηλεκτρικά. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τους μεγάλους καταναλωτές. Εκεί θα έχουμε αποτέλεσμα. Και κάτι που ε, δεν έχουμε στην Ευρώπη, έχουν στην Αμερική. Διαφοροποιημένες τιμές. Εδώ δεν υπάρχει κανένα, ε, κανένα κίνητρο. Γιατί αν το βράδυ 6 με 8 που είναι η μεγαλύτερη ζήτηση πληρώνω τα ίδια όπως τη νύχτα, ποιο θα είναι το κίνητρο που θα έχω να χρησιμοποιώ τη νύχτα τις συσκευέ μου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το διακανονισμό των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, να γίνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις ώρες εχμής και τις άλλες ώρες. Γιατί αυτό που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε τα δίκτυα και όχι να δώσουμε σε κάθε νοικοκυρό στην Ευρώπη κάποιο περίπλοκο μηχανηματάκι. Πρώτα, σε ευχαριστώ. Τρία λεπτά έχουμε ακόμα. Να δώσω το λόγο σύντομα στην Κομισιόν. Η κύριε Μουλονέ, ναι, αν προφέρω σωστά το όνομά σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια. Στο στάδιο αυτό, η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει την συγγήτρια για την πρωτοβουλία και την Επιτροπή. Συμφωνούμε με το πνεύμα των σχολείων που ακούσαμε τώρα. Ευχαριστώ. Dann gebe ich der Frau noch mal das Wort. Η κυρία Τόγια έχει βάλει το λόγο. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους ε, και ελπίζω και να υπάρξουν και άλλα σχόλια. Θα μοιράσω το σχέδιο της γνωμοδότησης για να διευκολύνω την ανταλλαγή των απόψεων ε, σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς ε, και να αναφερθώ σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για τους ευθύς μετρητές. Να επενθυμίσω ε, ότι η κυρία ΕΚ στην προηγούμενη θητεία είχε ε, καταθέσει ε, μια τροπολογία που ονομάστηκε βελτιστή πρακτική. Επίσης, ε, να σας πω ότι καθώς είμαι Ιταλίδα γνωρίζω πως έχει η κατάσταση και θα ήθελα να αρνηθώ το ότι αυτές οι προτάσεις έχουν εισαχθεί γιατί δεν καταβάλλονταν τα τέλη, δεν πληρώνουν την λογαριασμό. Κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό. Αλλά απλώς θέλαμε εδώ να διδάξουμε τους καταναλωτές τι χρησιμοποιούν. Δηλαδή ένας ευφύς μετρητής κάνει φύ και τον καταναλωτή να ξέρει τι χρησιμοποιεί και μάλιστα σε ορισμένε προσφορέ, ε, σε ορισμένε περιπτώσει απελευθέρωση, είχαμε και το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούνται συσκευέ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα συγκεκριμένο ωράριο. Εμείς ε, εδώ στην περίπτωση των οικοκυριών μιλάμε για τον αυτοέλεγχο της κατανάλωσης. Βέβαια έχουμε και την προβληματική των μεγάλων βιομηχανιών. Ευχαριστώ. Έκλεισε και η εξέταση αυτού. Τέλος της συνεδρίας λοιπόν σήμερα στην ώρα μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε κυρία Εκ να μιλήσετε. Ναι. Ναι. Εμείς ε, από την ομάδα των φιλελευθέρων ε, θέλουμε να συνεισφέρουμε τα μάλα σε αυτό το σημαντικό θέμα για το πώς θα ε, πετύχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και πώς ε, συστηματικά θα θεωρούμε τον τομέα των κτηρίων ε, και των μεταφορών ως ε, βασικούς τομείς και φυσικά μας ενδιαφέρει και το θέμα των φιών μετρητών και υπομονούμε να συνεργαστούμε. Πολύ ωραία. Πέρα λοιπόν τις συνεδρίασεις. Ακριβώς την ώρα μας θα αρχίσουμε τις συνεδρίασεις των τονιστών. Θα ήμουν ευγνώμων αν οι άλλοι συνάδελφοι βγαίνουν γλίγορα από την αίθουσα για να αρχίσουμε με ακρίβεια. Γιατί και εκεί δεν έχουμε υπερβολικά πολύ χρόνο. Μία ώρα που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.